Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Στάφαν Μιστούρα, τον οποίο και καλωσορίζω θερμά. Ο κύριος Στάφαν Μιστούρα είναι ο ειδικός απεστερμένο των Ηνωμένων Εθνών στη Συρία και μάλιστα είχε πολύ πλούσια εμπειρία στα Ηνωμένα Έθνη σε εμπόλεμες περιοχές. Ήταν και μάλιστα ε, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας. Κύριε Πρέσβη Μιστουρά, γνωρίζουμε ότι οι προσπάθειες για την εξασφάλιση ειρήνης και ε, σταθεροποίηση στη Συρία περνάνε από την ε, συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε πολλές ζώνες, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο συριακό πληθυσμό που έχει πληγεί από τις συνεχείς ε, σειράξεις και να επιτρέψει την ε, δρομολόγηση ανθρωπιστικής βοήθειας ειδικά σε ζώνες που ήταν ε, απρόσιτες εξαιτία των εχθροπραξιών. Και μάλιστα μία από τις ζώνες που θα μπορούσε να υποφεληθεί από τέτοια τοπική εκεχηρία θα είναι στο Χαλέπι το οποίο έγιναν σφοδρές μάχες για πολλούς μήνες. Έγιναν ε, επανειλημμένες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός στο Χαλέπι και την ανακήρυξη της ε, ελεύθερης πόλης για να αποφευθούν περαιτέρω αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Βέβαια υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Τι ρόλο θα έχουν τοπικές ε, συμφωνίες και σε, στη δημιουργία σταθερότητας και ασφάλειας στη Συρία, μια και ένα μεγάλο τμήμα της χώρας πλήττεται από τη βία και τη βαναυσότητα της, αυτο, της οργάνωσης που αυτοαποκαλείται Ισλαμικό κράτος. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και θα ήθελα να μας εξηγήσετε εξονυχιστικά τη χρήση των τοπικών συμφωνιών και χειρίες ως στρατηγική για την αποκατάσταση σταθερότητας και ασφάλειας στη Συρία. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε πώς θα εφαρμοστούν και θα διατηρηθούν τέτοιες συμφωνίες και χειρίες, τι ε, συνέπειες θα έχουν για τον τοπικό πληθυσμό και τι πολιτικές συνέπειες επίσης και αντίκτυπο θα έχουν. Είναι ε, ευαίσθητη αυτή τη στιγμή της πόλεμης ε, κατάστασης Συρία γιατί η Αίγυπτος και η Ρωσία προσπαθούν να αναβιώσουν το διάλογο και μάλιστα και το Ισλαμικό κράτος έχει τηθεί στο κομπάνι. Φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει η δυναμική, ακόμη και να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αποκατασταθεί ένας φυσιολογικός τρόπος ζωής στη χώρα. Παρακαλώ κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. E, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω αγγλικά, διότι είναι η πιο τεχνική γλώσσα που διαθέτουμε στα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, σουηδικά ή και γερμανικά ακόμα, είναι στη διάθεσή σας και μέχρι και αραβικά. Ε, ας αρχίσουμε όμως από τα αγγλικά με την άδεια σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας για τα θέματα που άπτονται της Συρίας. Σε σχέση με τα όσα μόλις είπατε, που είναι πάρα πολύ εύστοχα όλα αυτά που αναφέρατε, πρέπει να σας πω ότι με καθοδηγήσατε και για τον τρόπο που θα μπορούσα να διαρθρώσω τη σκέψη μου. Ε, μερικά γεγονότα, γιατί τα έχουμε ξεχάσει, έχουν τίνει να γίνονται στατιστικές. Διανύουμε το τέταρτο έτος του πολέμου στη Συρία. Είναι η στιγμή που έχουμε 12 εκατομμύρια ανάγκες, 7,6 εκατομμύρια εκτοπισμένοι, 2,3 εκατομμύρια πρόσφυγες, 200.000 εκτιμώνται, ίσως και περισσότεροι νεκροί, 1 εκατομμύριο Σύριοι ε, είναι τραυματίες. 4.000 σχολεία έχουν κλείσει, 219 αρχαιολογικοί, ιστορικοί τόποι και μνημεία είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερός είτε έχουν υποστεί ζημίες. Οποιοςδήποτε έχει πάει στη Συρία, όπως και εγώ και άλλοι από εσά σίγουρα, θα θυμάστε πόσο θαυμάσια καταπληκτική χώρα ήταν αυτή και θα παραμείνει ή θα ξαναγίνει. Αν κανείς πίστευε ότι θα μπορούσε να λυθεί η σύραξη στη η σύγκρουση με στρατιωτικά μέσα, ιδού η απόδειξη ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει λοιπόν στρατιωτική λύση. Αυτό το δέχονται οι πάντε, αρχίζει γενομένης από τον πρόεδρο Ασάτ και την κυβέρνησή του, μέχρι και την αντιπολίτευση και τι χώρες τη περιοχή και αλλού που ενέχονται ή ε, στο παρελθόν συμμετείχα. Όλοι έχουν ε, αναγνωρίσει ότι η λύση είναι μόνο πολιτική και λύση που θα την βρουν οι ίδιοι οι Στο μεταξύ, business as usual, σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα και είμαστε σε ένα τέλμα. Λες και όλα αυτά είναι απλή ρητορία, ενώ συνεχίζεται η σύραξη. Υπάρχουν όμως τα δύο εξή νέα φαινόμενα που έχουν αναδειθεί. Το πρώτο είναι η ανάδυση, οι δραστηριότητες στο Ιράκ και τη Συρία του ISIS, του Ισλαμικού κράτους. Και το άλλο γεγονός είναι η στρατιωτική αντίδραση από μια συμμαχία με επικεφαλής του Αμερικανούς για να αντικρουστεί αυτό, να αποκρουστεί. Κανονικά και παραδόξως θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε να λυθεί το πρόβλημα. Ε, καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος ε, βοήθησε να αναπτυχθεί το ISIS γιατί υπήρξε πρόσφορο και γόνιμο έδαφος επειδή υπήρχε κενό. Και εφόσον δεν νοεί τη στρατιωτική λύση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια πολιτική λύση. Τι έκαναν λοιπόν τα Ηνωμένα Έθνη και εγώ προσωπικά μέχρι τώρα, ποια ήταν η αποστολή μου. Από τους εξέχοντες προκατόχους μου και τον Κόφι Ανάν και τον Λαχτάρ Μπραήμι διδάχθηκα. Εκείνοι είχαν μια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση. Δηλαδή, σε ε, τεράστιες διεθνείς πρωτοβουλίες, μεγάλες διασκέψεις, έτσι ώστε να κοινοτοποιηθούν όσοι ενέχονται και τοπικός και διεθνώς για ένα πολιτικό διάλογο. Αλλά εξεδόθη ένα πολύ σημαντικό ε, ανακοινωθέν της Γενέβης, το οποίο είναι ακόμα σε ισχύ, Ταυτόχρονα έγιναν δύο διασκέψεις, οι οποίες όμως δεν έδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εμείς τώρα έχουμε διαφορετική προσέγγιση με τον ίδιο πάντα στόχο. Και ποια είναι η ιδέα. Ας επικεντρωθούμε τώρα στους εξή τρεις τομείς. Πρώτον, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειωθεί η βία. Βλέπουμε τα στοιχεία. Γιατί ο λαός της Συρίας αυτό ζητάει. Χαλάς, κυφάγια λένε στα αραβικά. Φτάνει πια, δεν αντέχουμε άλλο τέρμα οτιδήποτε μπορεί να βυθεί στην ανθρωπιστική βοήθεια για το λαό της Συρίας αυτή τη στιγμή μετά από τέσσερα χρόνια είναι κρίσιμο. Και είναι σε διασταυρούμενα πειρά. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε πλευρές τώρα έχουν και το ISIS. Ε, και είναι θύματα οι άνθρωποι και αυτό που θέλουν είναι να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Και αν εκεί υπάρξει οποιοδήποτε χώρος για ένα πολιτικό ορίζοντα, για ένα πολιτικό διάλογο μεταξύ των σύρων, θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία και να πιέσουμε. Και πάλι θεωρητικά όλοι συμφωνούν και τα θεωρούν λογικά όλα αυτά. Δεν είναι και πάρα πολύ φιλόδοξα, γιατί δεν μιλούμε για μια νέα Γενέβη 3, μιλάμε για βήματα συγκεκριμένα που πρέπει να γίνουν. Και δοκιμάσαμε να δούμε ε, τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό επιλέξαμε το Χαλέπι. Όλοι λέγουν και μου λένε ακόμα πολύ ότι τρελίστε. Το Χαλέπι είναι η πιο περίπλοκη περίπτωση. Είναι οι πάντες παρόντες εκεί οι αντιμαχόμενοι και κανείς δεν θα το δεχτεί. Με η απάντηση είναι ακριβώς επειδή είναι τόσο ε, ε, μεγάλη, δύσκολη περίπτωση, αλλά είναι το χαλέπι, είναι έμβλημα, είναι σύμβολο, είναι ένα κοκτέιλ όλων όσων υπάρχουν στη Συρία και ταυτόχρονα είναι ένα σύμβολο πόλη θρησκευτικού, ε, πόλη πολιτισμικού γίγνεσθε και είναι μια μεγάλη πόλη που δεν έχει πέσει στα χέρια της μιας ή της άλλης πλευράς. Και αν πέσει, 500.000 θα είναι οι πρόσφυγες προς την Τουρκία, ανθρωπιστική τραγωδία, πέρα από τα 3,2 εκατομμύρια των ήδη υφισταμένων προσφύγων. Και επίσης η πολιορκία είναι κατέρωθεν, γιατί χτυπιούνται ε, οι δύο πλευρές μέσα στην πόλη. Την τελευταία τριετία είναι μια μόνιμη πολιορκία. Γι' αυτό ε, κάναμε την πρόταση ε, να είναι όχι κατάπαυση του πυρός, γιατί η κατάπαυση του πύρος ε, στη Συρία δεν είναι κάτι το οποίο πείθει. Στη Χόμς και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες πόλεις είδαμε ε, ότι οι πόλεις είχαν καταρρεύσει και μας ζητούσαν τη βοήθειά μας. Ότι δεχόμαστε, συνθηκολογούμε, δεν, δεν πρόκειται γι' αυτό στο Χαλέπι, δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Ε, μιλάμε για πάγωμα ε, του μπαράζ ε, επιθέσεων, βομβαρδισμών από τη μια και από την άλλη όλμοι και οβίδες, αδιάκριτα και βροχίδων. Βεβαίως αναγνωρίζουμε ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι προτεραιότητα και όντως είναι και στη Συρία και στο Ιράκ. Βεβαίως αναγνωρίζουμε και κατονοούμε ότι στα ψηφίσματα 2170-2178 αντιμετωπίζουμε και θέματα της τρομοκρατίας που είναι η Αλνούστρα και το ΝΤΑΕΣ σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη και να σταματήσουν και οι ξένοι μαχητές ε, κατέρωθεν ή σε οποιαδήποτε πλευρά υπάρχουν αυτοί. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξουν κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τώρα για τα πολιτικά ζητήματα. Ε, εν ώψη όλων αυτών και επειδή είναι σε απόγνωση η κατάσταση, η ιδέα ήταν και παραμένει να φτιάξουμε ένα παράδειγμα. Να αρχίσει ο κόσμος να πιστεύει ότι υπάρχει κάποια ελπίδα για να μειωθεί η βία. Άρα να παγώσει η κατάσταση στο χαλέπι. Ε, ε, συζητούμε με τον Μπασάρ. Δεν είναι εύκολη η διαπραγμάτευση. Ξέρουμε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και αν δεν έχουμε μια ε, κατάπαυση του πυρός ε, κλασική παλαιομοδίτικη, αλλά ένα πάγωμα εκεί της κατάστασης, θα έχουμε δυσκολίες. Το χαλέπι είναι σαν το κομπάνι περίπου, ένα σύμβολο ε, που δείχνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να πέσει αυτή, αυτό το επίπεδο της βίας. Στο Κάιρο έγινε μια ε, συνεδρίαση, αλλά και στη Μόσχα και οι δύο μπορεί να μην είναι τέλειες. Για λόγους που αν θέλετε μπορώ να επεκταθώ. Αλλά εμείς τα υποστηρίξαμε. Γιατί οποιαδήποτε ευκαιρία παρουσιάζεται για πολιτικό διάλογο μεταξύ των σύρων, επαναλαμβάνω, έστω και με ατέλειες, έστω και με απουσίες, έστω και ε, αν είναι μερικοί από την αντιπολίτευση και κάποιοι από την κυβέρνηση, ό,τι και να είναι, είναι ε, καλύτερο βήμα από την, απουσία, την πλήρη απουσία διαλόγου. Και δεν υπάρχει ε, μηδενικό άθροισμα, δεν κερδίζει κανείς. Ε, μόνο χαμένους έχουμε σε αυτή την περίπτωση που είναι ο λαός της Συρίας. Άρα, ε, προγραμματίζουμε τώρα να συνεργαστούμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χρησιμοποιήσουμε το μοχλό που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη και τη δυνατότητα σύγκλησης για μια γενική συνολική προσέγγιση από σύσκεψη σε συνεδρίαση και να βρούμε κάποιο τρόπο, κάποια φόρμουλα. Δεν χρειάζεται να είσαι διαστημικός επιστήμονας για να τα βρεις αυτά. Υπάρχει πλαίσιο μετά τη Γενέβη, βεβαίως με προσαρμογή στη σημερινή πραγματικότητα, γιατί τότε στη Γενέβη δεν είχε αναδυθεί κόμμα το ΝΤΑΕΣ, ε, το ίσις, ε, αυτή είναι η αφετηρία όμως από την οποία μπορούμε να προχωρήσουμε και να ε, εργαστούμε. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε την αρχή, αλλά βρούμε ένα τύπο, ένα τρόπο, μία φόρμουλα για να μπουν όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Υπήρξαν προτάσεις, υφίστανται αυτές, ορισμένες είναι και πολύ ρεαλιστικές πρέπει να πω. Και τα πάντα ξεκίνησαν από μία έννοια. Να μειωθεί η βία, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και από εκεί και πέρα μπορείς να προχωρήσεις και στις συνταγματικές αλλαγές, και σε θεσμικές, η κυβέρνηση εθνικής ή πολιτική ενότητας, μετάβαση σε μια πολιτική κυβέρνηση που να συμμετέχουν όλες οι μειονότητες και η πλειονότητα φυσικά, οι πάντες στη Συρία. Και ενδεχομένως και εκλογές τελικά για να μπούμε σε μια διαφορετική κατάσταση. Δεν είναι ακόμα του παρόντος αυτό, θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι οι Σύριοι ε, έχουν εξαντληθεί. Και γενικότερα υπάρχει μια κόπωση. Δεν υπάρχουν νικητές, μόνο τρομερά δεινά, τρομακτικά. Τελευταίο σημείο, η Ευρώπη, εμείς, εσείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη εδώ και με παρηγορούν οι συνεδριάσεις που είχαμε τους 28 υπουργούς εξωτερικών της Ένωσης και την κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη πρόσφατα που απεκόμισα την αίσθηση ότι πάντες κατανοούν ότι έχει έρθει η ώρα της Ευρώπης να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή μέσω του ΙΕ δεν ξέρω μόνη της με κάποιο τρόπο να βρεθεί μια πρωτοβουλία για να σταθεροποιηθεί η Συρία. Και ένας τρόπος να γίνει αυτό, ακούω ότι γίνονται πολλές συζητήσεις, είναι ένα πακέτο, μία δέσμη ε, παρεμβάσεων, ας φανταστούμε πρώτα ο Θεός αν παγώσει το χαλέπι και γίνει αυτό που προτείνουμε μια ανοχήρωτη πόλη, ξαφνικά ε, τι βοήθεια θα δοθεί εκεί και άλλες πρωτοβουλίες έτσι ώστε ο κόσμος να καταλάβει τι τεράστιο πλεονέκτημα είναι αυτό και πόσο μεγάλη σπουδαία αλλαγή αν ακολουθήσουν όλοι ε, και όχι μόνο στο χαλέπι αλλά και παντού αλλού. Γι' αυτό ε, χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι εδώ. Σας ευγνωμονώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Μιστούρα, Μιστούρα, για τη Γενική Επισκόπηση που μας κάνετε. Ο κύριος Πλένκοβιτς ε, ζήτησε το λόγο. Ξεκινάμε την ε, ανταλλαγή απόψε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε μιστούρα σας ευχαριστώ θερμά για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Θυμάμαι τις δραστηριότητες σας πριν από 20 περίπου χρόνια και στην Κροατία και στη Βοσνία και Ριζεγοβίνη και πραγματικά έχετε πολύ πλούσια πείρα σε πολλές περιοχές του πλανήτη που χρειαζόταν διαχείριση κρίσεων. Είπατε ότι το Χαλέπι είναι, έχει συμβολικό χαρακτήρα και είδαμε ότι πάνω από 800 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Χαλέπι και 30 παιδιά. Μπορείτε λοιπόν να μας κάνετε μια εκτίμηση για την κατάσταση του καθεστώτος και της κυβέρνησης του Ασάντ. Γιατί ξέρουμε ότι το Χαλέπι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη, στα χέρια της αντιπολίτευσης. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι αξιόπιστο συνομιλητή ε, και τι πιθανότητε υπάρχουν ελπίδε για τη συνέχιση των συνομιλιών τη Γενέβη. Ευχαριστώ κύριο Σχόουιτ. Ευχαριστώ και σα είμαι ευγνώμων που ήρθατε κύριε Νταμιστούρα για να μα ε, παρουσιάσετε την κατάσταση και απόψει σα. Ε, έχετε την αμέριστη υποστήριξή μα. και θυμάμαι που είχατε δακρύσει όταν μας φορουσιάσετε την κατάσταση Σύρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πραγματικά ελπίζω να συνεχίσετε τις προσπάθειες και να μας, βρείτε, να μας βοηθήσετε να βρούμε κάποια λύση. Σας ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε για την μέχρι τώρα κατάσταση και είπατε ότι η πρόταση που βρίσκεται επιτάπητος δεν αφορά μια κατάπαυση του πυρός. Ο Υπουργός Εξωτερικών όμως του καθεστώτος του Μπασάρ Ελάσατ, είπε ότι είναι έτοιμοι να κάνουν στο Χαλέπι αυτό που έκαναν και στην πόλη Χόμς. Έτσι αντιλαμβάνεστε και εσείς τη θέση τους. Και από ό,τι κατάλαβα εγώ, η Συριακή κυβέρνηση έχει θέσει κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Την κατάθεση των όπλων εκ μέρους των, της αντιπολίτευσης, των ανταρτών. Κάτι που θα εμποδίσει πιστεύω την κατάληξη συμφωνίας. Πιστεύω ότι θα μπορείτε να υπερβείτε ε, αυτή την προϋπόθεση και την απέτηση που θέτει το καθεστώς του Πασάρ. Δεν μιλήσετε και τη θέση του Ιράν. Γιατί είπατε ότι πολλοί πιστεύουν ότι οι Χεσμολάχ του Ιράν θα βοηθήσουν ε, αντάρτες ε, ΣΥΙΤΕΣ να, να παίξουν σημαντικό ρόλο στις μάχες της Συρίας. Και την περασμένη εβδομάδα μάλιστα η παραστατική φρουρά του Ιράν είπε ότι η ηγέτης ε, του Ιράν έδωσε ε, διαταγή να ε, εφαρμοστεί και ένα πρόγραμμα για αποστολή και πυράβλων στο, στη Σύρια. Πιστεύετε ότι ο Ιράν θα επηρεάσει τη Σύρια, το επηρεάζει. Ποιες είναι οι ανησυχίες σχετικά τι κοινοποιείται αυτές τις ανησυχίες στο Ιράν. Και πιστεύετε ότι θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο από το Ασάντ ε, με το Ιράν και τι, ποια είναι η αντίδραση που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτό. Οι εκπρόσωποι του Μπασέρ Αλασάτ και τη αντιπολίτευση συμφώνησαν στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα να συνεχίσουν τι διαπραγματεύσει. Αλλά μέχρι στιγμή ε, δεν έχει βρεθεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια καινούργια στοιχεία, αν έχετε νέε πληροφορίε. Πάντω από ό,τι κατάλαβα η Συριακή Αντιπολίτευση επί του παρόντο τουλάχιστον δεν μπορεί να συμφωνήσει με τη ρωσική πρωτοβουλία. Και η μόνη συμφωνία αφορά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Πώς εκτιμάτε λοιπόν την κατάσταση. Πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα η αντιπολίτευση και ο εθνικός συνασπισμός της αντιπολίτευσης που είναι η πιο μετριοπαθή το πιο μετριοπαθή μέλη της αντιπολίτευσης να συμβάλλουν στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για να βρεθεί συμφωνία και τι προϋποθέσεις χρειάζονται για κάτι τέτοιο. Είναι αρκετό μακροσκελής ο κατάλογος των ομιλητών, γι' αυτό θα σας θερμοπαρακαλέσω να περιοριστείτε στο τρίλεπτο καθένας. Επειδή πολλοί σοσιαλιστές και δημοκράτες έχουν ζητήσει το λόγο, θα κάνω μια αναλλαγή των πολιτικών κομμάτων. Η κυρία Σάκε έχει το λόγο. Sorry, President, my name didn't come through as clearly. Δεν, δεν ε, άκουσα το, το όνομα μου. Είχατε τι γίνεται, έτσι γίνεται πολλές φορές με τα Ολλανδικά τα εκφωνούνται λάθο. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε αυτό το δύσκολο θέμα που οδήγησε σε τόσο σπουδαία άλλα ζητήματα σε σχέση με το τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρώπη ε, όσον αφορά αυτές τις απίστευτες ε, βαρβαρότητες και τον πόνο του Συριακού λαού, όπω θα τονίσατε κι εσεί. Επίση, μεγάλη μου χαρά που να μα μιλάτε για του ξένου μαγητέ και από τι δύο πλευρέ. Επομένω, ε, έχετε επίγνωση του ρόλου του Ιράν και των άλλων χωρών που έρχονται σε επικουρία. Τι εναλλακτικές έχουμε τόσο ώστε να σταματήσει αυτή η υπόθεση στη Συρία και τι σημαίνει αυτό για τον Άσαντ, για το ρόλο του. Άλλη ερώτηση. Έχουμε κάποια σενάρια σύμφωνα με το οποία εσείς θεωρείτε ότι οι διαπραγματεύσεις με ε, το Ισλαμικό κράτος είναι μια επιλογή, μια λύση. Τελευταία ερώτηση. Πώς θεωρείτε ότι συνδέεται η κατάσταση σε Ιράκ με την κατάσταση στην Συρία, όχι μόνο πλευράς ε, αιτίων. Γιατί είπατε και γι' αυτό το κενό εξουσία στη Συρία, είπατε ότι αυτό ε, περιέπλεξε την κατάσταση, αλλά επίση και ο πλευρά παραβλέπων συνεπειών όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση και όσον αφορά τα πολλαπλά μέτωπα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει κανεί για να καταστρέψει το ιστορικό κράτο και τι προκλήσει για την ευρύτερη περιοχή. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Πεγιόν, ο οποίο είναι ο εισηγητή μα ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να την ε, σταθερότητα και ασφάλεια στην ε, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Σε ευχαριστούμε που ήρθατε, λέει ο κ. Πέγιον. Ήταν πάρα πολύ εντελεχή η εισήγησή σα. Εγώ θα ήθελα αρχίζοντα να σα πω κάτι το οποίο καταλαβαίνω. Γιατί ισχύει για εσά ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Κάποιοι δυσαρεστήθηκαν με αυτό τότε που ο Ασάντ χρησιμοποίησε τα χημικά κατά του λαού του και χρησιμοποίησαμε αλλού τη στρατιωτική επέμβαση και πρέπει αυτό να το θυμόμαστε ότι υπάρχει μια στρατιωτική ε, συμμαχία με τις είπα οπότε αυτή είναι η αφετηρία τη τους του είπατε και επίσης όπως είπαν και οι συνάδελφοι τελικά δεν έχουμε ως επιλογή τη ερωτική επέμβαση ή όχι. Έχουμε όμως διπλωματική λύση ως, επιλογή. Άλλο τώρα. Αυτές οι διπλωματικές τις οποίες συζητούμε και μέχρι σήμερα παρά την γενική καλή θέληση ήρθαν σε αποτυχία. Μήπως είναι να δούμε σήμερα πού πηγαίνουμε και ακριβώς όπως ελέγχθη μια που θεωρείται ότι μπορεί να γίνει μια διάσκεψη για αφοπλισμό ή τέλος πάντων για συγκράτηση της βίας και των εχθροπαξιών και με τον Άσαν να πείσουμε όλες τις πλευρές ότι είναι εδώ να υπάρξει εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το λόγο κύριε Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε για την εισήγησή σας. Έχω τρεις ερωτήσεις. Είπατε για τις ε, συνομιλίες μέχρι τις 29 και είπατε για αυτές τις αρχές της Μόσχας και είπατε για όλα αυτά που μπορούν να συμφωνήσουν για την ενότητα της χώρας, να σταματήσουν τις πραξίες κλπ. Όμως είπαμε ότι ο επικεφαλής της ε, αντιπολίτευσης της ε, δεν συμμετέσχει. Μήπως θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να περιληφθεί σε αυτές τις ομιλίες και η συριακή θέση. Επίσης, είναι πάρα πολύ βασικός παίκτης στο Ισκακέρα και το Ιράν, το οποίο δεν συμμετέσχει στις συνομιλίες της Γενέβης. Υπάρχει περίπτωση να εμπλέξουμε το Ιράν σε διαπραγματεύσει στο μέλλον. Τέλος. Δικαιοσύνη, λογοδοσία, η ειρήνη. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να ξαναυπάρχουν στο προσκήνιο. Κάποιο είδους κάποιο είδου δικαστήριο επίση να υπάρξει για τη Συρία. Όμω, ε, εν ώψη του που κατέληξε τη διέξοδο το δικαστήριο τη Χάγη. Κύριε Μποργέση. Α, μιλάτε στο τηλέφωνο. Καλά, πάμε παρακάτω. Γκόμε. Α, μισό λεπτό. Α, μπορείτε να μιλήσετε. Ναι, βέβαια. Βέβαια, ευχαριστώ. Κύριε Μιστούρα, σας ευχαριστώ και εγώ. Κατά γνώμη μου, δεν φίξατε εις βάθος το θέμα των προσφύγων που ενδιαφέρει πολύ όσον αφορά τα σύνορά μας γιατί στο εξή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος τόσο ώστε να έχουμε κάποιο είδους ε, ε, είσοδο τρομοκρατών. Το επισημάνατε το πρόβλημα και όλα αυτά το οποία είπατε ενισχύουν την άποψή μας ότι υπάρχει κίνδυνος όπως έχουν πει ασχολούμενοι με την ασφάλεια. Τι μέτρα θα προτείνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο ώστε να υπάρχει συγκράτηση αυτού του κύματος μετανάστευσης και κάποια μέτρα ελέγχου. Να διαπιστωθεί επίσης το σε τι κίνδυνο βρίσκονται οι χριστιανικές μειονότητες της περιοχής διαφόρων επιμέρους δογμάτων. Και αυτό το έχουν πει πάρα πολύ έγκυροι. Και είχαμε εκκλήσεις, ούτως υπήρουν απελπισμένες προς την Ευρώπη. Τι διεθνής πρωτοβουλία προτίθεστε να αναλάβετε ούτως ώστε αυτό το πρόβλημα της δίωξης των χριστιανών της Ανατολής να γίνει θέμα προτεραιότητας όσον αφορά την πολιτική μας στις ε, παρέμβαση από πλευρά ε, ΟΗΕ και διεθνού κοινότητα συγκεκριμένα μέτρα. Όχι μόνο με διακηρύξει αρχή. Σα ευχαριστώ. Τώρα ήρθε η σειρά τη κυρία Γκόμε. Χαίρομαι που σα βλέπουμε κύριε Ντεμιστούρα. Η ερώτησή μου αφορά τη Συριακή Αντιπολίτευση. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα πήγαν στραβά και η εξέλιξη ήταν κακή επειδή ήταν κατακαιρματισμένη η Συριακή αντιπολίτευση. Δεν υπήρχε μια συμπαγής αντιπολίτευση στη Συρία. Υπάρχει τώρα κάποια μεγαλύτερη συνοχή. Υπάρχει πια μια εθνική πλατφόρμα που θα συνενώσει την αντιπολίτευση στη Συρία. Ε, βλέπετε κάτι τέτοιο να διαμορφώνεται εν ώψη των προσπαθειών που γίνονται στο Χαλέπι. Επίσης, σχέσεις ε, του Ισλαμικού κράτους με τον Ασάντ. Ε, το Ισλαμικό κράτος δεν είναι αντάρτε Σύριοι, δεν είναι τμήμα της Συριακής αντιπολίτευση. Είναι ένας ιδιότυπος συνασπισμό, άλλου είδου συνασπισμό, διεθνή συνασπισμό. Καμία σχέση με τον εθνικό συνασπισμό της αντιπολίτευση. Και μάλιστα στο Ιρακινό Κουρδιστάν ακούσαμε ότι υπάρχουν μερικέ περιπτώσει όπου ο Ασάντ συνεργάζεται με το Ισλαμικό κράτο με το ΙΣΙΣ. Εσείς τι πιστεύετε. Τέλος, ο ρόλος της Τουρκίας σε όλα αυτά. Έγινε μια προσπάθεια πριν από δύο χρόνια και μάλιστα εκεί διαδραμάτισε κέριο ρόλο η Τουρκία ε, και στήριξε τους ε, αντιφρονούντες στο Χαλέπι που μάχονταν κατά του ε, Ασάντ. Επίσης όμως είχαμε μια στήριξη της Τουρκίας που επέτρεψε την ε, προέλαση του ίσης στη Συρία και στο Ιράκ. Βέβαια, χρειαζόμαστε και την Τουρκία. Εσείς ε, τι γνώμη έχετε για όλα αυτά. Ωραία, τούρνο ε, Νάρ. Ο κύριος Νάρ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε και έχετε δίκιο ότι δεν έχει στρατιωτική λύση η σύγκρουση, αλλά η πολιτική λύση είναι λαβύρινθος. Πρώτον, διότι το ίσις είναι μια ε, ουσιαστική δύναμη εκεί και ασύμβατη με οποιαδήποτε ε, λύση μετά από διαπραγμάτευση. Δεύτερον, υπάρχει ένας κατακαιρματισμός ε, στην Συρία σε φυλές και σε θρησκείες και δόγματα. Οι αλαοίτες ε, κατέληξαν ε, να είναι σύμμαχοι των χριστιανών. Ίσως για τον ίδιο λόγο που ήταν σύμμαχοι με τον Σαντάμ Χουσέιν, γιατί δεν είχαν ιδεολογική συνάφεια μαζί του, αλλά θεωρούσαν ότι τους προστάτευε. Και έχουμε λοιπόν από τη μια τους χριστιανούς και κάποιους σουνίτες και απέναντι μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Και μεγάλη αντίφαση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ ε, είχαμε στο παρελθόν και των Αράβων και τώρα έχουμε αντίφαση μεταξύ των Αράβων των ίδιων στο εσωτερικό του αραβικού κόσμου. Και εσείς θεωρείτε ότι είναι αναπότρεπτη η παρουσία του Ιράν ως τμήμα της λύσης, της σύγκρουσης. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι και το Ιράν εκεί. Δεύτερον, εάν πραγματικά θεωρείτε, όπως και είναι η ειρηνική, η πολιτική λύση, ε, πώς θα λυθεί ε, το θέμα της δυναστείας των Αλάσατ δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι ένας άξονας ε, εξουσίας που συγκεντρώνει και κάπως συγκερνά τα διάφορα συμφέροντα των αλαοητών. Και πώς δύο θανάσιμοι εχθροί, όπως είναι οι αλαοίτες και οι χριστιανοί από τη μια και οι υπόλοιποι από την άλλη, θα μπορέσουν να συμφωνήσουν για να καταπολεμήσουν από κοινού το ίσις που είναι τόσο ακεραιόφρονες και ε, επειδή είναι τόσο φονταμεταλιστές, είναι ασύμβατοι, επαναλαμβάνουμε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Ο κύριος Σμιτ. Θα προσπαθήσω, Σμιθ, να μην επαναλάβω και άλλες ερωτήσεις. Κύριε Τεμιστούρα, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι όλοι εδώ σας υποστηρίζουμε και ακολουθούμε τις προσπάθειές σας με καθυσίχασε αυτό που αναφέρατε για την συνάντηση της Γενέβης και το κοινό ανακοινωθέν είναι η μόνη συμφωνία που υπάρχει σε αυτή τη μακρά περίοδο. Παραμένει στο κέντρο των προσπαθειών σας ε, ο σχηματισμός μιας μεταβατικής κυβέρνησης και βεβαίως θα πρέπει πρώτα να παγώσει ε, η η κατάσταση εκεί στο Χαλέπι, αλλά έχω τις αμφιβολίες μου και εσείς πιστεύω ε, δεν υπάρχει ο κίνδυνος όταν παγώσει η σύγκρουση σε διάφορες πόλεις μήπως μετατοπιστεί κάπου αλλού να το εκμεταλλευτεί δηλαδή αυτό η κυβέρνηση και κατά πόσο θα ε, συμμορφωθούν όλοι και ιδιαίτερα την πολίτευση και ποια, ποιο είναι το νομικό καθεστώς αυτών των ε, καταστάσεων και σε περίπτωση που κάποιος δεν συμμορφωθεί προς αυτό το πάγωμα των εχθροπασιών που το λέτε freeze και local freeze και όχι κατάπαυση του πυρός, πώς θα βεβαιωθείτε ότι θα συμμετέχουν και τι γίνεται με τους γείτονες Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ιράν για να υπάρχει μια ευρύτερη ε, συμμαχία και ένα συνασπισμός και όχι μόνο τοπική. Ο Κόρβιν Μίκε. Ε, thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Μιστούρα, θα ήθελα να σας πω ανοιχτά ότι κατά τη γνώμη μου δεν είστε πολιτικός. Εσείς ζείτε από τις συγκρούσεις. Άρα είναι προς το συμφέρον σας η σύγκρουση να κρατήσει όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί ε, είναι ο βιοπορισμός σας οι συγκρούσεις. Δεύτερον, μας είπατε ότι είναι αδύνατη μια στρατητική λύση. Μα πώς το ξέρετε. Μια παλιά παροιμία λέει ότι μπορεί όλοι να πιστεύουν ότι κάτι είναι απίθανο, κάποιος που έρχεται και δεν το πιστεύει ως απίθανο το κάνει και αλλάζουν τα πράγματα. Επίσης έχουμε τον ελεύθερο Συριακό στρατό. Ε, και αν μια στρατηγική, επιλέγαμε τη στρατηγική λύση, θα είχε ε, διορθωθεί το πρόβλημα εδώ και πολύ καιρό αν είχαμε στηρίξει τον ε, ελεύθερο Συριακό στρατό. Αλλά μόνο με συνομιλίε απλώς ε, θα παρατείνεται η σύγκρουση. Κοιτάξτε τη Τσετσενία. Ε, αιματηρότατη σύγκρουση, χειρότερη από τη Σύρια. Τώρα όμως ε, έχουμε άνθηση του κράτου τη Τσετσενία. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε μια ευκαιρία στην εξοχότητα του Μπάσερα Λασάτ. Ο κύριος Λίτς, παρακαλώ. Όχι, δεν ζήτησα το λόγο. Κυρία Σεμπάγιος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να πάμε πίσω το 2011 στην Αραβική Άνοιξη. Τότε που ο λαός της Συρίας είχε κατέβει στους δρόμους. Τι πήγε λάθο. Γιατί κατέληξε έτσι αυτή η κατάσταση. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, θα μπορούσαν οι γείτονε τη χώρα να κάνουν κάτι παραπάνω. Όταν όλα αυτά ξεκίνησαν στην Συρία, είχαμε ταυτόχρονα πόλεμο και στον Λίβανο. Στη Λιβύη. Και Μήπω θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι παραπάνω εκεί, στην αρχική φάση. Και τέλο πάντων να αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα, μαθήματα. Λιβύη και μετά Συρία. Να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επανεληφθούν αυτά. Θυμάμαι τότε, ήμουν μέλο του Ισουδικού Κοινοβουλίου και θυμάμαι ότι δεν προσέχαμε και πολύ τι γινόταν στη Συρία. Όλο για τη Λιβύη λέγαμε. Έγινε κάποια προσπάθεια να υπάρχει κάποια προσοχή και προστασία τη Συρία, αλλά δεν τα καταφέραμε γιατί τα στρατιωτικά ήταν πιο σημαντικά. Επομένω, ίσω μπορούμε τώρα να κάνουμε κάτι σε επίπεδο διπλωματία. Επομένω, μήπω θα μπορούσατε να μα πείτε σκέψει πάνω σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλέ ερωτήσει. Ο κύριο Σαφόζα. Σαφόζα. Έχετε τον λόγο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σύντομα. Ε, κύριε Πρέσβη, μας λέτε ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Και ο πρόεδρος άσε το ίδιο λέει. Άρα πώς θα προχωρήσουμε, ποιο είναι το πρόγραμμά σας, πιο συγκεκριμένα ερωτώ. Διότι βεβαίως αυτό είναι μια βάση συζήτησης, αλλά δεν μας βοηθάει να προοδεύσουμε. Δεύτερη ερώτηση. Συμφωνείτε ότι η υποστήριξή μας στη λεγόμενη δημοκρατική αντιπολίτευση ε, τελικά τις φετερίστηκαν κάποιοι, ο Ισλαμικός στρατός, Νταές, Ισής, όπως το λένε. Δηλαδή, το στρατιωτικό υλικό που στείλαμε εμείς στην ε, λεγόμενη υποτιθέμενη δημοκρατική αντιπολίτευση κατέληξε στα χέρια αυτών, στον Νταέ. Και επανέρχομαι στην ίδια ερώτηση που έκανε και η Άννα Γκόμες. Ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας. Τέταρτη ερώτηση. Εγώ ήμουν ε, πρόεδρος μιας οργάνωσης ε, στο νοσοκομείο του Χαλεπιού, η πρώτη μήκυο στην Σύρια. Εκεί πραγματικά έχουν συμμαχήσει οι Αλαουίτες και οι Χριστιανοί για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και πώς από αυτή την ενότητα μπορούμε να προχωρήσουμε για να επανέλθει και ενότητα γενικά στη χώρα. Πρακτικά, πώς το βλέπετε. Αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις είχα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ΙΕ για 1,5 δις απευθύνθηκε στην ε, διεθνή κοινότητα για να υπάρξει βοήθεια προς την Συρία. Λιγότερο από τα μισά βρέθηκαν. Η κατάσταση δε έγινε χειρότερη λόγω αυτών των βαρβαρικών ομάδων όπως το Ισλαμικό κράτος, τα χημικά από πλευρά του Άσαντ και επίσης ο κίνδυνος του να επεκταθεί η σύγκρουση σε Ιορδανία και Τουρκία. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια ειρηνική επίλυση του προβλήματος ε, κατόπιν της ανόδου ε, αυτών των ε, ακραίων ομάδων όπως είπαμε. Επίσης, για πετε μας ποιο πιστεύετε ότι είναι ο ρόλο του Ισραήλ σε αυτή την σύγκρουση. Πρόεδρος. Επόμενος, λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρέσβη που αναλάβατε αυτές τις δύσκολες προσπάθειες για αυτή την κρίση, λέει ο κύριος Φρόιντ. Πριν από λίγες μέρες ή μάλλον εβδομάδες είχαμε κάποιες ενδείξεις στροφής της Δύσης όσον αφορά την θέση τους προς τον Στην αρχή λέγανε ότι δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις μέχρι ότου παρετηθεί και αποχωρήσει. Τώρα όμως από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να μιλήσουμε μαζί του, θα πρέπει να τον συμπεριλάβουμε σε αυτήν την ανύπαρκτη την διαδικασία. Εσείς τι λέτε. Αυτό αυτή η στροφή. Διευκόλυνε το έργο σας ή το περιέβλεξε περισσότερο δεύτερο ερώτημα. Μη με παρεξηγείτε, αλλά είχαμε τον Κόφι Ανάν και, και, και άλλους ε, ε, εξαιρετικούς σας ε, προκατόφιου όπως τον Μπραχήμι επίσης και τι μπορείτε να κάνετε πώς θα διαφοροποιηθείτε σε σχέση με αυτούς τους πολύφερνους ούτως υπήν προκατόχους που δεν τα κατάφεραν όμως. Σειρά μου τώρα. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Μετά τις ε, ανησυχητικές ε, δράσεις που έγιναν στα ψήφιδα του Γολάν με την ε, επίθεση των Ισραηλινών και δυστυχώ είχαμε και το θάνατο ενό Ισπανού και ενόκρανου και δύο Ισραηλινών και μάλιστα εκφράσαμε τι ανησυχίε μα στην είπατε εκπρόσωπο γιατί ε, είχαμε και 11 ε, επιθεωρητές ε, του ΟΗΕ που ε, έπεσαν από τα Ισραηλινά πυρά γιατί δεν είχαν σταθερές θέσεις και τελικά έγιναν θύματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης προς το Λίβανο της σύγκρουσης αυτής, ε, γιατί έχουμε και τη πολλά που δραστηριοποιείται στη Συρία. Επίσης, αυτό το πάγωμα, το, το προσωρινό ή το τοπικό, που δεν είναι κατάποψη το πυρός, με Ποιο ήταν ο συνομιλητή σα, γιατί η ένοπλη αντιπολίτευση τη Συρία είναι πολύ μικρή και κυριαρχείται κυρίω από του τρομοκράτε του Ισλαμικού κράτου και άλλε ε, Ακραίε ομάδε εξτρεμιστικέ. Ποιο είναι το πρώτο βήμα για να συμπεριλάβουμε πολύ περισσότερους ε, τη αντιπολίτευση. γιατί ε, θα πρέπει να δούμε και τους ε, γειτονικέ χώρες που χρηματοδότησαν τη μία ή την άλλη πλευρά στην σύγκρουση. Ο κύριο Αγιάλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεμιστούρα γιατί είναι πραγματικά μια χτίδα φωτός ε, σε όλο αυτόν τον δρόμο και τη φρίκη που φαίνεται να είναι ατέρμονα. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για όλη την προσπάθεια που κάνει να βρει κάποια λύση. Είπατε ότι ο Συριακός λαός είναι εξουθενωμένος και γι' αυτό ακούγεται ότι πιο εύκολα θα ακούσουν μια πρόταση για πάγωμα της βίας. Και γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Συνήθως ε, ε, έχουμε κατάπαυση του πυρός σε τις περιπτώσεις, αλλά λέτε θα είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί μια κατάπαυση του πυρός. Εμείς όμως πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην πρόταση για το πάγωμα. Επίσης, ε, μιλήσατε για ένα άμεσο πακέτο ενίσχυσης, αρρωγής. Τι χρονοδιαγράμματα προβλέψατε με την κυρία Μογκερίνη, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εκεί για να βοηθήσουμε να εμπεδοθεί αυτή η κατάπαυση, το πάγωμα του πυρός. Μακάρι να πάει καλά η κατάσταση στο Χαλέπι και να γίνει υπόδειγμα και για τις άλλες πόλεις και για ολόκληρη τη Συρία. Να γίνει σύμβολο το Χαλέπι, ίσως για μια επαναφορά της κατάστασης προς μια μεγαλύτερη ομαλότητα. Ευχαριστώ. τώρα η ώρα και του κυρίου Ντεμιστούρα και πάλι. Δύσκολα τα βλέπω, δύσκολο το έργο του, γιατί πραγματικά τον υποβάλαμε σε ολόκληρη ανάκριση. Έχετε όσο χρόνο χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ. Μερικές ερωτήσεις ε, αλληλοεπικαλύπτονταν, αυτές θα τις ε, ομαδοποιήσω, άλλες όχι, γιατί ήταν πιο συγκεκριμένες και χρήζουν ξεχωριστής απάντησης. Θα προσπαθήσω πάντως. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ξεχωριστά σε κάθε ερώτηση και βοηθάτε με αν δεν καταφέρω να τα καλύψω όλα. Μπορούμε να... Μπορείτε να με υποθυμίσετε, επιθυμίστε αν κάτι, κάτι ξεχάσω. Στο Χαλέπι πρόσφατα είχαμε 100 νεκρούς, πριν από λίγες μέρες μόνο. Και μάλιστα από ρουκέτες της αντιπολίτευσης, όχι από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Και είχαμε από το μπαράζ των ε, Οβίδων ε, πολλούς αμάχους που έχασαν τη ζωή τους. Αλλά στο Χαλέπι ήταν από κυβερνητικές δυνάμεις οι Οβίδες και οι Όλμοι. Το Χαλέπι κατά το 2 τρίτα του ε, ελέγχεται από κυβερνητικές δυνάμεις. Μόνο το 1 τρίτο ελέγχει η αντιπολίτευση. Το Χαλέπι δεν ελέγχεται πλήρως από την αντιπολίτευση. Το αντίθετο συμβαίνει. Ένα μόνο μικρό τμήμα της πόλης ελέγχεται από την αντιπολίτευση. Και μάλιστα εμπλοκάρετε από ένα μικρό δρόμο. Και αν ε, ρίξετε μια ματιά σε αυτό το χάρτη, βέβαια μακριά σας είναι και δεν ξέρω αν βλέπετε καλά, κοιτάξτε τις ε, μαύρες περιοχές. Είναι η παρουσία του Ισλαμικού κράτους, του ISIS. Και πραγματικά ε, είναι συμβολική η θέση του Χαλέπ, του, της πόλης του Χαλεπιού και η κατάσταση είναι πραγματικά υπόδειγμα και δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή, σχεδόν ανέφικτη αποστολή, αλλά αν βρούμε μια λύση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο. Δύο τρίτα λοιπόν στι κυβερνητικέ δυνάμει βρίσκεται το Χαλέπι, ένα τρίτο στην αντιπολίτευση. Ένα τμήμα της αντιπολίτευσης είναι το μέτωπο Αλνούσρα που συντάσσεται με τους ε, τρομοκράτες και 20 χιλιόμετρα μακριά από το Χαλέπι βρίσκεται το ίσις, το Ισλαμικό κράτος. Έχουμε λοιπόν όλα τα συστατικά για να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση. Σκεφτείτε αν αναλάβει πλήρω τον έλεγχο η κυβέρνηση στο Χαλέπι. Μπορούμε να έχουμε 100.000 πρόσφυγες ε, που θα πρέπει να εξέλθουν από την ε, πόλη. Αν ε, το Ισλαμικό κράτος πολιορκήσει και ελέγξει την πόλη, θα έχουμε σφαγές και ίσως και 600.000 αμάχου που θα προσπαθήσουν να φύγουν ως πρόσφυγες. Και αν έχουμε μαζικό βομβαρδισμό από την κυβέρνηση, θα κατασπαραχθεί η πόλη. Και αν είχε πάει κανεί στο Χαλέπι, γνωρίζει ποια είναι η συμβολική αξία αυτής της πόλης για τη Συρία ολόκληρη. Και αν ήσασταν μαζί μου στο Χόμς, όπως που πήγα πρόσφατα, θα το καταλαβαίνετε. 43 χρόνια παρακολούθησα 21 συγκρούσει. Πήγα και στο Ντουμπροβνίκ. Πήγα σε πολλέ εμβόλεμε ζώνε με φρίκη και τρόμα, πουθενά δεν είδα κάτι παρόμοιο με αυτό που είδα στο Χόμς πλήρως ε, κατεστραμμένο και μια νεκρή πόλη. Αυτό ήταν πραγματικά ανευπροηγουμένο. Θα πρέπει να βρούμε, ε, βρούμε μια λύση για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο για το Χαλέπι. Περίπλοκη κατάσταση και η δολοφονία 100 αμάχων την πριν από λίγε μέρε είναι απόδειξη ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι όσο δύσκολη και είναι η κατάσταση. Τώρα, οι παρενέργειες που χρησιμοποιούμε στους στρατιωτικούς και οι παράπλευρες απώλειες, είναι πραγματικά πολύ δύσκολος όρος στρατιωτικός. Το Χαλέπ είναι το ίδιο συμβολικό όσο και το κομπάνι. Θυμάστε, κανένα δεν ήθελε να επέμβει και υπήρχαν πολλοί, πολλοί λόγοι για να μην γίνει τίποτα και το κουομπάνι είχε ακόμη κρατήσει. Ουσιαστικά μια γυναίκα κράτησε την αντίσταση. Και το Χαλέπι έγινε τώρα διεθνώς ζήτημα και αυτή η διεθνής προσοχή απέστηκε τουλάχιστον την κατάρρευση της ε, πόλης που την περιμέναμε σχεδόν το Δεκέμβρη. Δεν έγινε η τελική μάχη στο Χαλέπι και έτσι κράτησε η πόλη αυτή. Βέβαια, ακριβώ επειδή είδαμε ότι χάθηκαν πρόσφατα 100 άμαχοι, είναι ένα επιπλέον λόγο για να επικεντρώσουμε τι προσπάθειέ μα. Τώρα, οι προποθέσει για τις συνομιλίες για το Χαλέπι. Όντως, η κυβέρνηση της Συρίας, όταν υπέβαλε την πρόταση για το πάγωμα των εχθροπραξιών στο Χαλέπι, άρχισε να θέτει όρους, προϋποθέσεις, όπως αναφέρατε. Είπατε, οι ξένοι μαχητές να εγκαταλείψουν ε, την χώρα ή να ε, μπουν στον Συριακό στρατό ή να αφοπλιστούν, να καταθέσουν τα όπλα τους ή να αναγνωρίσουν την ε, ενότητα της πόλης και τον έλεγχο τον κυβερνητικό στην πόλη. Θεωρητικά είναι εύλογες αυτές οι αρχές και είναι αλήθεια ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να εγκαταλείψουν την Συρία οι ξένοι μαχητές και αργά ή γρήγορα θα πρέπει να εξαλειφθεί η παρουσία των τρομοκρατών στη Σύρια. Τα ψηφίσματα 2170 και 2178. Κάποια στιγμή πρέπει να επανενωθεί η Συρία και όχι να διαιρεθεί. Κανένα δεν προτείνει κάτι που να διαιρεί τη Συρία. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να τεθεί ω προπόθεση για να σταματήσουν οι εχθροπραξίε, τουλάχιστον στη χρήση βαρέων όπλων ε, στο Χαλέπι. Εξαρτάται πώ θα το θέσει κανεί. Ω προπόθεση ή ω πιθανή συνέπεια μετά από μια συμφωνία. Γιατί όλοι συμφωνούμε. Δεν θέλουμε ξένους μαχητές, δεν θέλουμε τρομοκράτες, μια ενωμένη χώρα και μια ενιαία κυβέρνηση που θα εξασφαλίζει τον έλεγχο ολόκληρη της χώρας και θα αποκαταστήσει τη σταθερότητα. Οπότε συνεχίζονται οι συζητήσεις, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα, κανένας δεν περίμενε από την κυβέρνηση να ενδώσει και να υποχωρήσει σε βασικά σημεία της, αλλά θα συνεχίσουμε, δεν θα εγκαταλείψουμε το χαλέπι. Ιράν τώρα. Το Ιράν είναι πολύ σημαντικό. Η επιρροή του είναι σαφής, η παρουσία του σαφής. Η Χεσμολάχ ε, βάρινε στις μάχες και έκανε τη διαφορά. Πριν από λίγους μήνες φαινόταν ότι κέρδιζε η αντιπολίτευση. Υπήρξε όμως μια σημαντική αλλαγή επιτόπου. Και κατά τη γνώμη των αναλυτών αυτή η στροφή οφείλεται και στην ανάμειξη της Χεσμολάχ. Τώρα θέλουμε ανάμεξη του Ιράν σε μια λύση για τη Συρία. Αναμφισβήτητα, ναι. Γιατί χωρίς το Ιράν, χωρίς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς την Τουρκία, χωρίς ανάμεξη αυτών, αυτών των χωρών και συμμετοχή τους σε μία φόρμουλα, χωρίς τη Ρωσία, χωρίς τις Ηνωμένε Πολιτείε, χωρίς τα κράτη της περιοχής, δεν θα δημιουργήσουμε την απαραίτητη κρίσιμη μάζα για να φέρουμε κάποιες αλλαγές και εξέλιξη στη Συρία. Και σίγουρα με ανάμεξη και του Ιράν, με συμμετοχή και του Ιράν. Κατά τη γνώμη μου η συμφωνία ήταν αγαστή πρωτοβουλία γιατί η κυβέρνηση της Ρωσίας έχει επιρροή και βαραίνει ο λόγος της στη, στη Συρία, στην κυβέρνηση της Συρίας και η πρωτοβουλία που ανέλαβε και η προσπάθεια που έκανε να φέρει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και την ε, Συριακή κυβέρνηση είναι πολύ σημαντική γιατί θέλουμε την Συριακή κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις για να ξεκινήσουμε τις ε, δύσκολες συζητήσεις για το τι εστί κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, χωρίς προϋποθέσεις και με συμμετοχή όλων. Δεν είναι καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο. Και το γεγονός ότι στη συνάντηση απουσίαζε εκπρόσωπος επίσημος ε, της ε, Συριακής Αντιπολίτευσης και αποσίαζαν και σημαντικοί αντιφρονούντες όπως ο Αλχατίπ, σίγουρα δεν είναι καλό σημάδι. Αυτό όμως που συνέβη στη Μόσχα, η συνάντηση της Μόσχας ήταν ενδιαφέρον και χρήσιμο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Είχαμε 11 σημεία από τη συνάντηση, μερικά θα τα συζητήσουμε, μερικά ε, είναι συναφή και πλησιάζουν και το ανακοινωθέν της Γενέβης. Προτιμούμε οποιαδήποτε εξέλιξη από μια παθητική, ε, μυρολατρική, το συμπεριφορά που λέμε να περιμένουμε το τέλος ε, της ε, σύραξης και μετά να έχουμε άλλο 300.000 θύματα. Και να πάω στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να σας πω ότι λυπούμε, είχαμε απώλειες 300.000 και απευθύνουμε έκκληση σε όλους να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να επανέλθουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Business as usual. Κάιρο και Μόσχα όχι τέλειες συμφωνίες, συνομιλίες, αλλά χρήσιμες. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με την ε, στήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Οτιδήποτε όθηση και πρόοδος σημειωθεί είναι ευπρόσδεκτη. Τώρα τι μπορείτε να κάνετε εσείς, ήδη έχετε κάνει πολλά ε, και χαίρομαι που το ξαναρωτήσατε. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βοηθήσει τις προσπάθειές μας. Θα ήταν ε, σίγουρα ευάρεστο να πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν νοείται στρατιωτική λύση, όπως έχει αναγνωριστεί. Και να παγώσουν οι εχθροπραξίες, οι μάχες στο Χαλέπ. Αυτό να το πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το λέω αυτό γιατί μέσω αυτής της δήλωσης θα δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα για να μην έχουμε μετά από ένα τρίμηνο, τετράμινο ε, ένα ακόμη στατιστικό στοιχείο στο Χαλέπι όπως έγινε και με το κομπάνι να χρησιμοποιήσουμε και το Χαλέπι ως συμβολική πόλη ως σύμβολο και να πούμε ό,τι και να κάνετε υπάρχουν και όρια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο ένα χρόνο και να έχουμε άλλους 300.000 ε, νεκρούς. Ο ρόλος του Μπασάρας Αλασάντ για το μέλλον. Αυτό εγώ θα το άφηνα να το κρίνει και να ασχοληθεί ο Συριακός Λαός. Η δε πρόταση για πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποια κυβέρνηση συνασπισμού όπου θα συμμετέσχουν όλοι και όταν λέω όλοι εννοώ όλοι χριστιανοί, αλαουίτες, Κούρδοι, ε, Δρούζοι όλοι όλοι και βεβαίως η σουνητική πλειοψηφία το πρόβλημα είναι και ότι έχουν ε, εξαιρεθεί όχι βέβαια οι Ισλαμικό κράτος γιατί δεν θέλουν και έτσι να οδηγηθούμε σε κάποια ανθεώρηση του συντάγματος που χρειάζεται και στη συνέχεια να πάμε σε εκλογές. Και σε τι δεν θα τους περιλάβει όλους, γιατί ο, ο Άσαντ εκπροσωπεί 50% του πολιτισμού, τόσο όταν τους ελέγχει. Σχεδόν το μένα της χώρας ελέγχει και σημαντικό τμήμα της χώρας. Δεν μπορώ το αγνοήσουμε αυτό μετά από μια τετραετία που ε, είδαμε ότι όλα τα υπόλοιπα οδηγούν σε αδιέξοδο. Πάντως αυτή η διαδικασία θα πρέπει να οδηγήσει σε μια διαμόρφωση της πολιτικής ε, συγκυρίας που να είναι σταθεροποιητική. Όλοι να περιλαμβάνουν τώρα διαπραγματεύσεις με το ζωικό κράτο. Με τίποτα. Ούτε ούτε θα κάνουν στο τραπέζι με εμάς. ούτε εμείς στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Είναι τρομοκράτε. Έχουν χαρακτηριστεί επισήμως από τον ΟΗΕ. Παρ' όλα αυτά, έχω σφίξει το χέρι του Σαντάμ Χουσέιν, του Μιλόσεβιτς, του Νατζιμπουλάχ και είναι πολλοί από αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκράτε και το έκανα αυτό και δεν μπορώ να σας πω ότι η μαμά μου θα ήταν περήφανη για αυτό που έκανα αλλά χρειάστηκε να συζητήσω μαζί τους κάποιο είδου ανθρωπιστική βοήθεια για τον κόσμο που αυτοί ήλεγχαν τότε που ήλεγχαν κάποιο χώρο. Οπότε από ανθρωπιστικής πλευράς νομίζω ότι ο, ο ΙΕ πάντοτε θα πρέπει να είναι έτοιμος να κάτσει στο τραπέζι με οποιονδήποτε για να μπορέσει να αγγίξει με κάποια ανθρωπιστική κίνηση τον κόσμο, όχι από πολιτική πλευρά. Δεν συζητούμε, δεν δραματευόμαστε. Είναι οργάνωση τρομοκρατική. Το μόνο το οποίο να κάνουν είναι αυτά που πρόσφατα έχουν κάνει. Και σας ευχαριστώ. Τώρα, σχέση Ιράκ με Συρία. Ε, είναι προφανές ότι υπάρχει σχέση. Μα γιατί ίσως δεν έχει ούτε σύνορα σε πολλά σημεία μεταξύ των δύο χωρών. Και ο ίδιος έχω εργαστεί προηγουμένως στο Ιράκ και θυμούμαι πάρα πολύ καλά ότι αυτό που σήμερα ονομάζουμε Ισλαμικό κράτος, ίσως τέλος πάντων, τότε ήταν ο Ζαρκάουι και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι τότε εκμεταλλεύτηκαν το διέξοδο, την απογοήτευση των Σουνιτών που είχαν μείνει απ' έξω από όλες τι εξελίξεις από το Γκάμιντ και κατόπιν και στο Ιράκ. Την κυβέρνηση τέλο πάντων. Και ε, κατόπιν είχαμε την Αλκάιντα. Ε, πήραν τα πράγματα την κατεύθυνσή του. Ήταν πολλά, πολλά λάθη και έτσι πήγαμε στη Συρία και τώρα ξαναγυρίζουμε στο πρόβλημα του Ιράκ. Φυσικά και είναι αλληλένδετα τα προβλήματα και θα πρέπει επομένω και τα δύο να τα αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα και παράλληλα τα μιλούμε ιδίω για το Ισλαμικό κράτο τώρα. Αστάθεια στη Συρία, ναι, δημιούργησε αστάθεια στο Ιράκ, αλλά και ισχύει και το αντίστροφο. Τώρα, εάν εμπιστευόμαστε τον Άσαντ σε επιτρέψει που κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μα το μεγαλύτερο πρόβλημα σε τέτοιε φάσει είναι ακριβώ η έλλειψη εμπιστοσύνη. Ε, κανείς δεν πιστεύεται κανένα άλλο. Και κάποια στιγμή ελπίζω θα μπορέσουμε να έχουμε συνομιλίες. Γιατί κανένας, ούτε ο Λάσαντ, ούτε η αντιπολίτευση μπορεί μόνος του να προχωρήσει. Άρα χρειάζεται η αρρωγή όλων ημών, ακριβώ όπως έχει γίνει και σε άλλες συγκρούσεις. Και έτσι να μπορέσουμε όλους να τους ε, ε, εξωθήσουμε να κάτσουν και να δουν ένα γίνοντιο μέλλον για τη Συρία, η Μόσχα. Ναι, και η αντιπολίτευση θα μπορούσε να ασχοληθεί. Αν υπήρχε όμως εμπιστοσύνη και υπήρξε κάποια ευκαιρία που χάθηκε. Εάν σταματούσαν οι συγκρούσεις στο Χαλέπι και αν αυτό ήταν πρόσφορά της η κυβέρνηση τέλος πάντων, τότε νομίζω ότι πολλοί από την αντιπολίτευση θα ενδιαφερόντουσαν να συμμετάσχουν. Έτσι θα θεωρούσαν ότι είναι κίνηση αυτό για δημιουργία εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση, ούτω ώστε να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον για μείωση των εχθροπραξιών. Οπότε, να πια είναι η ευκαιρία να διευρυνθεί ο συνασπισμό. Αυτοί που θεωρούν ότι χρειάζεται διάλογος ε, ακόμα και με τον εχθρό. Πρόσφυγες. Είναι τραγικό το πρόβλημα. Μίλαγα τις προάλλες στη Γενέβη των Αντώνιο Κουτιέρες Πολύ περισσότεροι είναι τώρα οι πρόσφυγες από την ε, Συρία παρά οι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν. Έχω πάει δύο φορές στην πόστολη στο Αφγανιστάν και πρέπει να σας πω ότι εγώ θεώρησα εκεί ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, είναι πάρα πολύ αυτή. Α, τώρα όμω είπαμε είναι πολύ περισσότεροι και φυσικά αποσταθεροποιούν τι χώρε. Για φανταστείτε, μια μικρή χώρα σαν τον Λίβανο, και εκεί έχω εργαστεί. Ε, είναι σαν να είχαν, είπα, 100 εκατομμύρια πρόσφυγε σήμερα. Για φανταστείτε, τι θα οι είπα. Είναι το αντίστοιχο, αναλογικά, το ότι ε, έχει αυτές χώρε από του, από τη Συρία πιο από όσους έχουν έρθει από την Παλαιστίνη ως πρόσφυγες. Βέβαια, όπως είπε ο κ. Μπορκέσιο, δεν έχω να πω πολλά σε σχέση με το ότι εκεί στα στρατόπεδα των προσφύγων έχουμε διείσδυση πολλών ε, από πλευράς του Ισλαμικού κράτους. Πάντως, ε, η μόνη περίπτωση κατά την οποία εγώ το διαπίστωσα αυτό να γίνεται είναι στον Λίβανο, από την Αλνούσουρα. Και αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα για το ιστορικό της χώρας. Και όπως ξέρετε, ε, και αυτό έχει οδηγήσει από σταθεροποίηση του Λιβανού. Βεβαίως όμως και θα πρέπει να παρακολουθήσουν την κατάσταση. Η δε μεγάλη πλειοψηφία των προσφύγων από την ε, Συρία ε, υφίστανται κάποιους ε, ελέγχους ε, και φύγανε γιατί φοβόντουσαν την κυβέρνηση. Πάντως οι περισσότεροι απλώς είναι πρόσφυγες ταπεινωμένοι, φοβισμένοι, ήταν ε, περήφανοι άνθρωποι, αλλά τώρα ταπεινώθηκαν και περιμένουν πότε θα τελειώσει ο πόλεμος να πάνε στη χώρα τους. Περισσότεροι από αυτούς έχουν ε, ε, σπουδάσει και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα καμία δουλειά τώρα παρά μόνο να περιμένουν. Τώρα σαν αυτές τις διώξεις των χριστιανών και των μειονοτήτων θα προσέθετα σε Ιράκ και Συρία. Αυτό είναι ένα ε, μεγάλο πρόβλημα και οποιαδήποτε ε, λύση δοθεί θα πρέπει να καλύψει και αυτό το πρόβλημα. Το Ισλαμικό κράτος είναι η βασική μας μέρη, η βασική μας ανησυχία. Αλλά βέβαια και η νόσορα έχει κατηγορηθεί ότι έχει καταστρέψει εκκλησίες και έχει διώξει χριστιανούς, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να ε, μείνουμε το μόνο μέλλον για τη Συρία είναι το να αγκαλιαστούν όλοι, όλοι να περιληφθούν, να μην μείνει κανείς απ' έξω. Αυτή τη στιγμή ε, ανησυχούν και οι χριστιανοί και οι αλαουίτες. Ε, γι' αυτό και θα πρέπει να τους καθησυχάσει η διεθνής κοινότητα και ο ΙΕ. Όταν δε θα βρεθεί μια πολιτική φόρμουλα, τότε θα σταματήσουν οι διώξεις. Θα συμπεριληφθούν στη λύση αυτή. Να, τώρα για την Λιβύη, όπως είπατε, καλά τα είπατε θα πρέπει να αντιλήσουμε συμπεράσματα. Να ωφεληθούμε από τα λάθη του παρελθόντος κάθε φορά που συζητούμε για την Συρία με οποιονδήποτε, όλοι μου υπενθυμίζουν. Ας αποφύγουμε αυτό το οποίο έγινε στην Λιβύη. Να το αποφύγουμε εξασφαλίζοντας ότι θα εξευρεθεί το νωρίτερο δυνατόν πολιτική λύση. Δεν ήμουν εκεί βέβαια, δεν μπορώ να σας πω τι έγινε και τι δεν έγινε τότε Εάν τότε στη Λιβύη είχαμε φροντίσει για μια γρήγορη πολιτική λύση, δεν θα υπήρχε Ισλαμικό κράτος, δεν θα υπήρχε διείσδυση των ε, ξένων μαχητών και από τις δύο πλευρές. Κάνοντας τώρα τόσο δύσκολο να πάμε σε διαπραγματεύσεις. Σωστά είπατε. Ακόμα και για το Χαλέπι. Πρέπει κανείς τώρα να κάτσει και να συζητήσει όχι με δύο ή τρεις ομάδες, με 18. Κάποια στιγμή η ιστορία θα τα κρίνει αυτά γιατί όντως χάθηκαν ευκαιρίες και θα πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Έχω υπηρετήσει στο Ιράκ και θυμάμαι πάρα πολύ καλά και όλοι αυτό το παρεδέχτησαν ότι το μεγαλύτερο λάθος ήταν το ότι διαλύσαμε τους θεσμούς, τα θεσμικά όργανα, το στρατό. Πάρα πολύ τώρα που είναι στο Ισλαμικό και πριν ε, ανήκαν στην πρωτική φορά του Ιράκ. Άρα το μυστικό και είναι αυτό το οποίο όλοι το παραδέχονται και, και το λέει και το ανακοινωθέτη της Γενέβης είναι ότι ό,τι και να γίνει στη Συρία τα θεσμικά όργανα ή θεσμοί και ο στρατός θα πρέπει να διατηρηθούν και να προστατευτούν τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποιο είδους κατάρρευση ακριβώς όπως έγινε και στο Ιράκ και ακόμα χειρότερα ότι έγινε στην Λιβύη. πώς θα μεγαλύτερη συνοχή στην αντιπολίτευση. Μα αυτό ελπίζουμε και ελπίζουμε να το ελπίζουν και οι ίδιοι. Το πρόβλημα είναι ότι τους υποστηρίζουν διάφοροι περιφερειακοί παίκτες εκεί, δυνάμεις που ε, δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα. Εκπροσωπούν συμφέροντα άλλων περιφερειακών δυνάμεων περισσότερο και λιγότερο τα ίδια τους τα συμφέροντα και τώρα έχουν καταλάβει όλο και περισσότερο ότι θα πρέπει να δείξουν ότι δεν είναι αδύναμοι. Και στο Κάιρο είχαμε κάποια εθαρρυντικά σημεία και μηνύματα. Είναι σημαντικό, γιατί όταν συναντάτε και την κυβέρνηση σου λέει δεν έχω συνομιλητή. Έχω κάτι γκρουπούσκουλα εκεί πέρα, αντί να έχω μια αντιπολίτευση συντεταγμένη απέναντί μου. Άρα είναι σημαντικό και για μας για να καταλάβουμε ότι μιλούμε με κάποιον που είναι ένας συνομιλητής αξιόπιστος αλλά και συνεπής. Ε, σιγά σιγά έχω την αίσθηση ότι προς τα εκεί πηγαίνουν αλλά θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε και να τους οθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ο ρόλος της Τουρκίας. Καταρχάς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μια χώρα που έχει 900 χιλιόμετρα σύνορα πάνω κάτω με το ίσις, Ιράκ και Συρία και 1,6 εκατομμύρια πρόσφυγες είναι μια χώρα η οποία επλήγει πάρα πολύ από τις συνέπειες και φοβάται ενδεχομένως και νέες συνέπειες. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε και τις δικές τους ανησυχίες σε ό,τι αφορά τον ρόλο τους για κάτι δημοσιεύματα που είδαν ε, το φως και που είπατε κι εσείς, εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι η Τουρκία παραγνωρίζει τα ψηφίσματα, τα γνωρίζει πολύ καλά, 2170 και 2178. Δηλαδή, να μην βοηθούμε καμία μετακίνηση ξένων μαχητών και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει βοήθεια τρομοκρατικής ομάδας. Δεν έχω λόγους να πιστεύω ότι ισχύει το αντίθετο. Αλλά θα πρέπει και επί τόπου η Τουρκία να αποδεικνύει ότι ανησυχεί. Ανησυχεί μήπως τις έρθουν και άλλες 400.000 πρόσφυγες. Από πού? Από το Χαλέπι ακριβώς καταρρεύσει και αυτή η πόλη. Περιφερειακές δυνάμεις, πολύ σημαντικό. Όταν συζητούμε για το Ιράν δεν θα πρέπει να λησμονούμε πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε και τη θέση της Σαουδικής Αραβίας και άλλων μιζώνων δυνάμεων εκεί που ανησύχησαν πάρα πολύ από την κατάσταση ε, στη Συρία οι Σουνίτες που είναι πλειονότητα έχουν πληγεί πάρα πολύ από τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, ενώ στην αρχή ήταν πολύ ειρηνική εξέγερση ας πούμε και κατέληξε σε αυτή τη βία και οδήγησε και σε τρομακτικές ε, φρικαλαιότητες. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα. Πώς μπορούμε να φανταστούμε αλαουίτες, χριστιανούς και σουνίτες να συνεργάζονται Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος σε μια χώρα σαν τη Συρία όπου ήταν ε, δεδομένη η συμβίωση, αλλά βέβαια με ανισορροπίες μεταξύ των κοινοτήτων και θα πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν νοείται τίποτα διαφορετικό. Στο κάτω-κάτω κοιτάξτε το Λίβανο. Είναι ένα τεράστιο ψηφιδωτό ε, αλλά έχει μια αξιοθαύμαστη δυνατότητα επιβίωσης παρά το γεγονός ότι είναι πολλές διαφορετικές κοινότητες από τους Μαρονίτες αρχής γενομένης μέχρι τη Χεσμολά. Αλλά βρήκαν ένα τρόπο συμβίωσης με τις ατέλειές του, αλλά είναι αξιοθαύμαστος. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τις δυνατότητες των σύρων, αν δεν εμπλέκονται διεθνείς ε, παράγοντες που πιέζουν για στρατιωτικό αποτέλεσμα και από πολλέ πλευρέ, από όλε τις γίνεται αυτό. Α του αφήσουμε να καθίσουν οι Σύριοι να βρουν μια Συριακή λύση. Όπω βρήκανε και οι Λιβανέζοι με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών και τη διεθνού κοινότητα, αλλά η λύση ήρθε από το Λίβανο. Ποια είναι η εναλλακτική ε, λύση χάο στην περιοχή Λίβανο, Τουρκία, Ιορδανία, κατάρρευση τη Συρία και παρουσία του Ισλαμικού κράτου στι ακτέ τη Μεσογείου. Για την ε, βοήθεια που στείλαμε στην αντιπολίτευση αν κατέληξε στα χέρια του ίσης είναι πιθανότατο διότι κάποιοι από την αντιπολίτευση τελικά ε, υποκλήθηκαν στην άλλη ρούστρα και στο Ισλαμικό κράτος. Ξαφνικά βρέθηκε ο που είχε δοθεί σε μια ομάδα της αντιπολίψησης που θεωρεί το μετριοπαθής έπεσαν στα χέρια του Ισλαμικού κράτους. Αλλά τα περισσότερα όπλα που έχουν ε, ήταν στη Μοσούλη. 85.000 ε, ε, στρατιωτικοί εξαφανίστηκαν. Άφησαν τα όπλα τους και 4-4.500 μαχητές του Ισλαμικού κράτους μπήκαν στη Μοσούλη και έχουν αρκετή όπλισμό για να συνεχίσουν ένα ε, μακρύ πόλεμο και μάλιστα υψίστης τεχνολογίας ε, όπλα. Ε, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες και έχουν μεγάλες ποσότητες και μεγάλα οικονομικά αφού έπεσε στα χέρια του η Μοσούλη. Είναι εκπληκτικά αυτά και πάλι για τους Αλαούτες και τους ε, Χριστιανούς. Προχτές κάποιος στη Δαμασκό είπε, ένας Άραβας, Σουνίτης, και πολύ σωστά είπε ότι το μέλλον της νομιμοποίησης οποιασδήποτε κυβέρνησης είναι σε δύο λέξεις μέσα, συμπερίληψη και ανάπτυξη, ένταξη. Και οι Σουνίτες, Σιήτες, Κούρδοι, Αλαούιτες, Χριστιανοί, χωρίς αποκλισμούς, Αλλιώς εκεί δεν θα χωράει ούτε το ε, Ντάις, ούτε το Ισλαμικό κράτος, ούτε κανείς για να παίζει το χαρτί της τρομοκρατίας και να υποδίεται ότι έτσι θα λυθεί ένα τέτοιο πρόβλημα. Θυμηθείτε ότι ένα από τα σφάλματα που βγήκαν από τη διάσκεψη της Βόνης για το Αφγανιστάν ήταν ότι είχαν αποκλειστεί οι τιμένοι. Οι παστούν είχαν υποεκπροσώπηση και δεν ήταν κανονική η παρουσία τους. Πράγμα που τους έκανε ευάλωτους προς τους Ταλιμπάν που τους πήραν στην αγκαλιά τους και τους είπανε ορίστε εμεί θα υπερασπιστούμε τα δικά σας συμφέροντα. Αυτή η φόρμουλα ε, σας αποκλείει. Έτσι τους φέρουμε στο πιάτο, σε ένα σημαίνιο δίσκο, τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουν και να το κεφαλαιοποιήσουν αυτό το γεγονός. Έγινε μια πολύ ειλικρινή ερώτηση προς εμένα, κύριε. Έχετε δίκιο. Πώς μπορώ να φανταστώ. Άνθρωποι που θεωρώ ότι είναι άξιοι και άριστοι διαπραγματευτές. Ο Κόφι Ανάν, βραβείο Νόμπελ και σπουδαίος γενικός γραμματέας και ο Λάχτερ Ιμπραχήμι που ήταν ο εμπνευστής και μέτρα διαφόρων λύσεων, εγώ πώς είναι δυνατόν να τους ε, διαδεχθώ και να κάνω κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν έχω καμιά εγγύηση για το αποτέλεσμα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι μετά από 43 χρόνια στον ΟΗΕ σε 21 περιοχές εμπόλεμες και με σειράξεις, το μόνο που ξέρω είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη ε, δεν έχουν την πολυτέλεια να θεωρούν ε, ότι ε, δεν έχει σημασία η παρουσία τους και να τα, ε, ε, το βάλουν κάτω και στη Σεμπρένιτσα και στη Ρουάντα και παντού. Εάν μου πείτε ότι είναι επικίνδυνη αδύνατη αποστολή και θα πρέπει να ε, σηκώσω τα χέρια ψηλά, δεν θα συμφωνήσω. Δεν ξέρω αν θα κάνω τη διαφορά, θα προσπαθήσω. Βεβαίως σε κάθε κρίση υπάρχει και μια ευκαιρία. Και όταν ανέλαβα αυτή την αποστολή μετά από 43 χρόνια, η μόνη αίσθηση που είχα ήταν ότι το Ισλαμικό κράτος ε, και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση είναι μια φρικτή κρίση αλλά μπορεί να είναι και ευκαιρία για όλους για να κινητοποιηθούν και οι Σύριοι και οι εκτός Συρίας και όσοι κάνουν εκεί πολέμους δι' Ε, αφήνουν ε, την χώρα ε, ενδεχομένως στα χέρια ενός τέρατος. Μιλήσατε για την Τσετσενία, για την Ρωσία και για άλλους. Μπορούμε εμείς αυτή την αποτρόπαια εξέλιξη να τη χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία αν παγώσει, ας πούμε, παγώνει ε, η σύραξη στο Χαλέπι. Σταματάνε τις ομοβροντίες πυρών οι δύο πλευρές. Και πολεμάει μόνο το Ισλαμικό κράτος. Θα ήταν πολύ εύκολο η Διεθνή Συμμαχία να επικεντρωθεί ε, σε αυτούς που θέλουν να καταλάβουν όλη την περιοχή. Αν έχεις εκεί διάφορες ομάδες που διτίθεται και πολεμάνε μία την άλλη, τότε θα έρθει το Ισλαμικό κράτος σαν ένα τεράστιο μαύρο πουλί από πάνω και θα ε, επιτεθεί ε, ως αρπακτικό όταν θα έχει οριμάσει η κατάσταση. Θα μπορούσε η σύγκρουση λέτε να μεταδοθεί στο Λίβανο. Βεβαίως υπάρχουν ε, τέτοια μηνύματα και μόνο χάρη στην αξιοθαύμαστη στάση των Λιβανέζων και των πολιτικών αυτό πετράπει το συζήτησα με τον Πρωθυπουργό και πρόσφατα διαπίστωσα ότι υπήρξαν ε, στιγμές που ήταν στο παραπέντε. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτό, αλλά η λύση και πάλι για να αποφευθεί είναι να λυθεί στη Συρία το πρόβλημα, για να μην μεταδοθεί. Το πακέτο πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοήθησε. Αν πετύχει στο Χαλέπι, ναι, χρειάζεται να δοθούν κάποια κίνητρα στον κόσμο και στο Χαλέπι και αλλού για να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια ελπίδα εάν παγώσει εκεί η σύγκρουση. Εάν δεν παγώσει, στο Χαλέπι καθυστερήσει, μπορούμε να το εφαρμόσουμε και σε άλλες πόλεις. Γιατί ο λαός έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει. Είναι εξουθενωμένοι μπορούν να πούν και στην Αλνούστρα δεν συμφωνείς με το πάγωμα, αλλά αν αρχίσεις τώρα ε, να ε, πυροβολείς ενώ όλοι οι άλλοι έχουν σταματήσει, εσύ ε, έχει σταματήσει τα τρόφιμα και το γάλα που περιμένουμε για τα παιδιά μας και η Αλνούστρα δεν μπορεί, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια να το κάνει. Συμπέρασμα, δεν υπάρχει πανάκια, ε, το ξέρω ότι είναι επικίνδυνη η αδύνατη αποστολή, αλλά πρέπει να την αναλάβουμε. Στους Financial Times ήταν, ένα πολύ αστείο άρθρο που έλεγε ότι ε, οι πιο επικίνδυνες δουλειές στον κόσμο σήμερα και δύσκολες είναι οι εξή. Και η δική μου θέση ήταν ε, η παρήθμου 6. Και η 7η ήταν ο κουρέας του Κίμιλ Σούγκ. Η αμέσως επόμενη σε επικινδυνότητα. Ε, είναι περίπλοκη λοιπόν η κατάσταση, αλλά δεν ε, έχουμε την πολυτέλεια να την ε, παρατήσουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για την πολύ διαφωτιστική αυτή ενημέρωση που μας κάνατε και που απαντήσατε διεξοδικά σε όλες τις ερωτήσεις. Επίσης θα ήθελα να σας συγχαρώ και για κάτι άλλο. Στην Επιτροπή μας συχνά έχουμε πολύ ε, σφοδρές και αρνητικές πολλές φορέ συζητήσει. Αυτή τη, αυτή τη φορά είχαμε μια πολύ θετική ε, ομιλία, πολύ αισιόδοξη που δεν επιχείρη καθόλου να κάνει κατήχηση η χειραγώγη. Σας ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα για την παρουσία σας και την ομιλία σας. Μια μικρή διακοπή μέχρι τις 5.30. Ευχαριστώ. Vamos Συνεχίζουμε. Το τμήμα αυτό προβλέπει κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Έχω εξεβονίμων την κυρία Λίδα Μάκαβαν που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης και συμπρόεδρος ε, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψε με τον Γιάννη Ελίασον, που είναι αναπληρωτή ε, Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Αθηνών. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον καλεσμένο μα, τον κύριο Γιάννη Ελίασον. Περιμένω λίγο για να βάλει τα ακουστικά του. Καλωσορίζω θερμά τον κύριο Γιάννη Ελίασον, που είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Αθηνών. Και είναι μεγάλη τιμή για μας Λίγο ησυχία παρακαλώ. Τιμή για μας που επισκέπτεται ο κύριος Ελίασον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να λάβει μέρος σε αυτήν την κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τον κύριο Μαϊν Χάρτινγκ, που είναι πρέσβη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έχουν στενή συνεργασία σε θεσμικό επίπεδο, που μάλιστα τα τελευταία χρόνια εντατικοποιήθηκε, ιδιαίτερα στι προσπάθειε ε, εμπέδωση τη ειρήνη και διαχείριση κρίσεων οι δύο κοινοβουλευτικές μας επιτροπές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και προσβλέπουν σε μια ευρύτερη και βαθύτερη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών. Πρόσφατα, ο ΙΕ ξεκίνησε διάφορες πρωτοβουλίες και το 2015 θα έχει αποφασιστική σημασία για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η πλήρης αναθεώρηση των ειρηνευτικών αποστολών με επικεφαλή τον κ. Σραμό Σόρτα και οι αποστολές διατήρηση ειρήνης αλλά και οι πολιτικές αποστολέ. Η εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Και τέλος, το πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015 και το πρόγραμμα για τις κλιματικές αλλαγές είναι πολύ σημαντικά θέματα. Το 2015 ε, ο ΙΕ θα χαράξει τη μελλοντική του πορεία και φυσικά θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, τις εξελίξεις στον οργανισμό αυτό. Κύριε Ελίασον, ε, θα ήθελα να μας, πείτε, να μας παρουσιάσετε τη γνώμη σας για αυτές τις ε, μείζονες προκλήσεις που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ο ΙΕ και πώς θα το κάνει. Μας ενδιαφέρει επίσης η γνώμη σας ε, για την ε, σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία και κάποιες προτάσεις ίσως για να συγκεκριμενοποιήσουμε και την πολιτική μας στο θέμα αυτό. Πρώτα μας θα δώσω το λόγο στην Συμπρόεδρο, την κυρία Λίντα Μάκαβαν, που όπως είπα είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Εξωτερικών και Ανάπτυξης. Εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης, ε, στην οποία προεδρεύω, θα ήθελα να εστερνιστώ τις παρατηρήσεις του κυρίου Κόουσου και να σας καλωσορίσω θερμά στη σημερινή μας συνεδρίαση, γιατί τα θέματα που σας απασχολούν είναι εξαιρετικά σημαντικά όχι μόνο για τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών, αλλά και για τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης και ο κύριος Μάι Χάρτινγκ, ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη είναι παρόν και θα ήθελα να καλωσορίσω και εκείνον θερμά. Όπως είπε ο κύριος Κόουσο, το 2015 θα είναι ορόσημο για τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί συνεχίζονται πολλές διαδικασίες ε, τις οποίες παρακολουθούμε εκ του και εμείς. Το Μάρτιο θα λάβει χώρα η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών ε, για την ε, Ιαπωνία και για, την, για τις φυσικές καταστροφές εκεί και θα έχουμε και την, ε, τον Ιούλιο για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των κρίσεων και επίσης το Σεπτέμβριο τη Σύνοδο Κορυφής για την αντικατάσταση των στόχων της χιλιετίας και των βιώσιμων στόχων της χιλιετία. θέμα αυτό μα απασχολεί ιδιαίτερα και έχουμε στενές συνεργασίε με του συναδέλφου από την Ηνωμένα Έθνη. Και τέλο το Δεκέμβριο θα γίνει στο Παρίσι η διάσκεψη ε, κορυφή για τι κλιματικέ αλλαγέ. Κάτι που θα χαράξει τη, την πορεία της αναπτυξιακής πολιτικής για το μέλλον. Και μάλιστα και για μας το 2015 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε ποια είναι τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναπτυξιακή πολιτική, τι προέκυψε από τη διαδικασία των στόχων της χιλιετίας, αλλά να δραστηριοποιηθούμε και να αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες και να προωθήσουμε νέο πρόγραμμα για τη νέα ε, αναπτυξιακή μας ατζέντα. Εσείς, ε, ως αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θα προωθήσετε τις αντίστοιχες προσπάθειες του ΟΗΕ και σίγουρα είναι σημαντική η χρονιά αυτή και για τον οργανισμό σας. Περιμένουμε λοιπόν με αδημονία την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Συμπρόεδρε, κυρία Μάκαβαν. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την πρόσκληση που μου κάνατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές είναι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών και μάλιστα εκπροσωπείται μια οργάνωση που είναι πολύ σημαντικός παγκόσμιος φορέας και παράγων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην ε, αποκατάσταση ειρήνης ε, και ασφάλειας, αλλά και στην ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θα επικεντρωθώ σε αυτούς τους τρεις τομείς, λοιπόν, ε, κύριοι συμπρόεδροι, με την άδειά σας. Νομίζω ότι σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο όπου δοκιμάζει τους παγκόσμιους οργανισμούς και την πολυμέρεια, αλλά και τους εθνικούς ε, θεσμούς και θεσμικά όργανα. Θα πρέπει λοιπόν να ικανοποιήσουμε την παγκόσμια κοινή γνώμη, τις προσδοκίες της για ασφάλεια, αλλά και για ανάπτυξη, για ειρήνη και για ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι η αξιοπιστία αυτών των θεσμικών οργάνων ε, που δημιουργήθηκαν για την ευημερία των πολιτών. Έχω πάντα στην τσέπη μου το χάρτη το Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το 1982. Είναι η 12η εκδοχή της Χάρτας ε, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Ας θυμηθούμε τις τρεις πρώτες λέξεις αυτής της χάρτας. Εμείς οι λαοί. Αυτές είναι οι πρώτες τρεις ε, λέξεις, γιατί αυτούς τους λαούς υπηρετούμε. Και νομίζω ότι αυτό, αυτή θα είναι και η ίστατη πράξη λογοδοσίας και ανάληψη ευθύνης εκ μέρους των οργανισμών μας. Αυτή η αλλαγή του τοπίου που πραγματικά αλλάζει ραγδαία και μεταλλάσσεται καθημερινά, έχουμε νέα στοιχεία της γεωπολιτικής και γεωοικονομικής κατάστασης. Έχουμε έκρηξη των τεχνολογιών ε, επικοινωνίας και πληροφορίας, έχουμε όλο και αυξανόμενο ρόλο της μετανάστευσης, ε, της αστιφιλίας, Δυστυχώ και άνοδο της τρομοκρατίας σε συνδυασμό με το οργανωμένο έγκλημα. Τεράστιες είναι οι προκλήσει ε, που έχουμε ενώπιον μα και τεράστιες οι ευθύνε να τις ε, αναλάβουμε και να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες των, Ευρω... των παγκόσμιων πολιτών. Βέβαια δεν έχουμε μόνο ζωφερές ειδήσει. Ε, πολύ ενθαρρυντικό στην παγκόσμια σκηνή είναι ο όλο και μεγαλύτερο ρόλος των γυναικών και επιτέλους αρχίζουν και παίρνουν οι γυναίκες τη θέση που θα, θα έπρεπε να είχαν πάρει εδώ και πολύ καιρό. Τώρα, για το πρόγραμμά μας. Όταν ήμουν πρόεδρος ε, της ε, Γενικής Συνέλευσης, ε, ξελέγει το 2005, διαμορφώσαμε το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών με τρόπο που φαντάζομαι θα το δεχτείτε και εσείς. Δηλαδή, δεν νοείται ειρήνη χωρίς ανάπτυξη και δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς ειρήνη και τίποτα από τα παραπάνω δεν νοείται χωρίς σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρόσθεται και το κράτος δικαίου. Αυτά είναι τρία ελληλέδετα τμήματα του, των διεθνών προτεραιοτήτων. Αν ένας από τους πυλώνες ε, είναι ασθενής, ολόκληρο το οικοδόμημα κλονίζεται. Και το είδαμε και επί τόπου. Τι σημαίνει όταν ε, ο πόλεμος υπονομεύει την ανάπτυξη και οι καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταπατούν, ε, μάλλον κλονίζουν τη συνοχή των κοινωνιών. Θα πρέπει ταυτόχρονα να συντρέχουν και οι τρει προϋποθέσεις Και όχι διαδοχικά. Όταν ήμουν μαθητή, ένας καθηγητή μου είπε πρώτα έχουμε την ανάπτυξη. Ή μάλλον πρώτα έχουμε την ειρήνη. Μετά την ανάπτυξη και μετά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι, λάθος. Θα πρέπει ταυτόχρονα να προωθούμε και τις τρεις έννοιες. Είναι συνειφασμένες ε, μεταξύ τους. Και βλέπω τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Σλοβακίας, τον κύριο να ε, συνεργαστήκαμε στενά για το θέμα αυτό στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, η σημαντικότερη πρόκληση στο θέμα της ε, ασφάλειας και της ειρήνης, είναι κάτι που το συζητάτε και εδώ, είναι η Συρία. Δεν θα επεκταθώ γιατί ο Στάφαν Ντεμίστουρα ήρθε προηγουμένως και σας ενημέρωσε είναι σαν μόλιση στο σώμα, στο παγκόσμιο σώμα ε, αυτή η κατάσταση. Καταστράφηκε ε, το έθνος, ε, δυνοπάθησαν οι πολίτες της Συρίας. Οι πρόσφυγες υπονομεύουν την ασφάλεια και την ευημερία των γειτονικών χωρών. Πήγα στο Λίβανο πριν από ένα μήνα και ένας στους τέσσερις κατοίκους του Λιβάνου είναι από τη Συρία σήμερα. Πήγα και στη Βηρητό. Οι μισοί μαθητές σε ένα σχολείο της Βηρητού είναι Σύριοι. Για να αφήσουμε την πίεση στα σχολεία, στη δημόσια υγεία, στην απασχόληση είναι προφανή. Και είδαμε και τα αποτελέσματα της κρίσης της Συρίας στο Ιράκ με την άνοδο της τρομοκρατίας και την επέλεση και επέκταση του Ισλαμικού κράτους. Ε, θέλουμε ψήφισμα του ΟΗΕ και ο Λάχταρ Μπραχίμη και ο προκατοχός του Κόφι Ανάν προσπάθησαν να πολύ σκληρά, αλλά πραγματικά δεν είχα την απαραίτητη μυϊκή δύναμη, το σφρίγος για να κάνουν αυτό που έπρεπε. Προσπαθήσαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον τις ανθρωπιστικές συνέπειες τεράστια διαστάσεων με τεράστια κρίση προσφύγων αλλά και τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Πέραν τούτου έχουμε και την κρίση στη, στην Αφρική. Και θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό παράδειγμα που θα μπορούσα να αντιλήσω από την κρίση στην Αφρική είναι ότι θα πρέπει να τη δούμε αυτή στο περιφερειακό πλαίσιο. Ήμουν στον Ταρφούρα διαμεσολαβητής του 2008 και μετά από μήνες που ήμουν διαμεσολαβητής, από ένα μήνα κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μόνος μου δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Ούτε στο, μόνο στο Σουδάν. Έπρεπε να πω στο Τσάντ, στη Λιβύη, στην Ερυθρέα για να βρω λύση και για να φέρω τις εμπλεκόμενες πλευρές στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και την αντιπολίτευση στον Ταρφούρ και στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, θα πρέπει να δούμε τις κρίσεις στο περιφερειακό πλαίσιο. Τη Συρία στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο Κονγκό για παράδειγμα, έχουμε μια κατάσταση που μόνο όταν διευρύθηκε η, το, η ατζέντα του ΟΗΕ και πέρασε και στο πολιτικό πλαίσιο και ξεπέρασε το πλαίσιο της ειρήνης, μόνο τότε όταν διευρυθήκαμε και στο πολιτικό σκέλος σημειώσαμε κάποια πρόοδο. Και όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, ένα σημαντικό σύννεφο εδώ είναι τα αυξανόμενα προβλήματα που μας δημιουργεί η κρίση στην Ουκρανία. Δεν σας κρύβω ότι το όλο διεθνές κλίμα επιδεινώθηκε από αυτή την κατάσταση και φαίνεται ότι αρχίζει και ε, μας ξαναφοβίζει το φάντασμα του ψυχρού πολέμου. Θα πρέπει όμως να περιορίσουμε τις ζημιές που είναι ήδη πάρα πολλές. Καταρχήν ε, έλλειψη εμπιστοσύνης είναι προφανές, αλλά υπάρχει κίνδυνος ε, να επεκταθεί αυτή η σύγκρουση και σε άλλες περιοχές. Χρειαζόμαστε συνεργασία, όπως ε, και στη Συρία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, για να μην μιλήσουμε για τις σημαντικές διαπραγματεύσεις 5 συν 1 για το Ιράν. Θα πρέπει επίσης ε, να μείνουμε αμετάκλητοι και αδιάλεκτοι στην τήρηση των αρχών του, διεθνούς δικαίου σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση που θα έχει ανυπολόγιστες και καταστροφικές συνέπειες. Άλλο σημαντικό θέμα που ενδιαφέρει κυρίως την πρόεδρο Μάκαβαν είναι η ανάπτυξη, ο δεύτερο πυλώνα. Και θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό έργο που έχουμε στα Ηνωμένα Έθνη για το δεύτερο πυλώνα είναι το έργο για τους στόχους της νέας γενιάς ε, που θα καταρτιστούν από το τέλη Σεπτεμβρίου. Ξέρετε ότι 8 από τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας ε, ανταποκρίθηκαν στο, στο σκοπό τους και θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο τώρα της, του στόχου της εκρίζωσης της φτώχειας. Αλλά έχουμε πολύ σημαντικό έργο, όχι μόνο για την εξάλληψη της φτώχειας, αλλά και για τη βιωσιμότητα. Και η πρώτη φορά είναι που πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο για την υγεία του πλανήτη, αλλά για το μέλλον του πλανήτη. Γιατί στη ζωή μπορεί να έχουμε δεύτερο εναλλακτικό σχέδιο, αλλά σίγουρα δεν έχουμε εναλλακτικό πλανήτη για να μετακομίσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε το στόχο της εξάλληψης της φτώχειας με την βιωσιμότητα, το στόχο της αηφορίας. Από εδώ και πέρα την αηφορία θα πρέπει να τη συμπεριλάβουμε σε όλους μας τους στόχους. Επίσης, ε, και το κράτος δικαίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, η σημασία των θεσμών για την ανάπτυξη. Και μάλιστα κατάγομαι από μια χώρα, τη Σουηδία, που κάποτε ήταν από τις φτωχότερες στην Ευρώπη, με άλλες σκανδιναβικές χώρες. Τελικά μεταξελίχθηκε σε μια πολύ ευημερούσα χώρα και κοινωνία και εν μέρη χάρη στις επενδύσεις, στις υποδομές, στην παιδεία και σε καλούς θεσμούς. Και νομίζω ότι αυτό είναι κέρια σημασία για να καταπολεμήσουμε την φτώχεια και να έχουμε ένα υφόρο μέλλον. Χρειαζόμαστε θεσμούς που θα εξασφαλίζουν τη συνέχεια των προσπαθειών μα. Για τι διαπραγματεύσει λοιπόν αυτέ έχουμε πολλέ προκλήσεις και θα έλεγα ότι η πρωταρχική πρόκληση είναι να βρούμε καλέ λύσει για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξη. Γιατί στο G77 πολλέ χώρε Ασία, Λατινική Αμερική και Αφρική λένε ότι Έχουμε πολλά καλά χρηματοδοτικά προγράμματα για τις κλιματικές αλλαγές, αλλά σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης δεν βλέπουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, συγκεκριμένα νούμερα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτή την πρόκληση. Στα μέσα Ιουλίου θα γίνει σχετική διάσκεψη κορυφής και εκεί θα δούμε αν μπορούμε όντως να βρούμε λύση στο θέμα της χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα γιατί υπάρχει το επιχείρημα που λέει οι επενδύσεις στις κλιματικές αλλαγές ισοδυναμούν σήμερα με τις επενδύσεις στην εξάλληψη της φτώχειας. Όντως ισχύει κάτι τέτοιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σίγουρα συμβάλλουν. Αλλά θα πρέπει να βρούμε και νέους τρόπους χρηματοδότησης, νέα μέσα χρηματοδότησης. Και πιο συνήθιστους ε, τρόπους ε, για να χρηματοδοτήσουμε την ε, ανάπτυξη. Πέραν τη επίσημη ενίσχυση για την ανάπτυξη, που ελπίζουμε να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο, να δούμε τα συνταξιδοτικά ταμεία στον ιδιωτικό τομέα, ε, κινητοποίηση εθνικών πόρων ή παράνομη ροή χρηματοδότηση. Ο πρώην πρόεδρο τη Νοτιού ο Ταμπόι Μπίκη, είναι επικεφαλή μια ομάδα που κατέληξε στο συμπέρασμα με επιστημονικά πορίσματα, με αδιάστατα τεκμήρια, ότι 50 δισεκατομμύρια δολάρια φεύγουν παράνομα από την Αφρική κάθε χρόνο. Αν μπορέσουμε να επαναπατρίσουμε αυτά τα χρήματα, σίγουρα είναι σημαντική πηγή χρηματοδότηση. Επίσης, το θέμα της άφεση του χρέους, της διαγραφής του χρέους ή της απομείωσης του χρέους. Και το θέμα το, της φορολογίας ή μάλλον της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων που είναι ένα τμήμα της ευρύτερης εικόνας. Και τα λέω όλα αυτά γιατί είναι σημαντικό ήδη από τώρα, γιατί είμαστε Φεβρουάριο και έχουμε την συζήτηση τον Ιούλιο, θα πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί ε, δεν θα προλάβουμε αν δεν κινητοποιηθούμε μέχρι το τέλη Σεπτεμβρίου να ελοπίσουμε τους στόχους. Και ένα τελευταίο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το καλοκαίρι του 2013 ο Γενικός Γραμματέας Μπάνκι Μουν και ο υποφαινόμενος λάβαμε μία έκθεση από συναδέλφους που ε, είδαν ε, τα τελευταία στάδια του πολέμου στη Σρι Λάνκα και τη μελέτησαν και κατέληξαν στο πόρισμα ε, ότι τα Ηνωμένα Έθνη κρίθηκαν ένοχα γιατί συστηματικά δεν κατάφεραν να διαγνώσουν τι συνέβαινε εκεί. Και είδαμε το πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πρώτη γραμμή για να αναβαθμιστεί ο ρόλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός ε, των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει λοιπόν εμείς οι λαοί να δίνουμε αξιοπρεπή ζωή στους άλλους λαούς και να σταθούμε στο ύψος ε, της οικουμενικής διακήρυξης. Έτσι θα κάνουμε στο μέλλον, δεν πρόκειται να περιμένουμε να γίνουν και φρικαλαιότητες ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα κάνουμε τη φωνή μας να ακούγεται περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και στο Συμβούλιο Ασφαλείας και θα επισημαίνουμε καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε φρικαλαιότητες ακόμα και σε εθνοκάθαρση και ε, γενοκτονία. Κάθε φορά που είπαμε ποτέ πια κάτι το ξαναείδαμε και είχαμε αποτυχία επί αποτυχίας. Αυτό θα πρέπει να τερματιστεί. Εγώ δεν λέω ότι στο μέλλον αυτά θα αποφεύγονται, αλλά τουλάχιστον να κατανοήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι η παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η πρώτη σεισμική δόνηση ε, προειδοποιητική που θα πρέπει να την ακούμε. Και γνωρίζω ότι το κοινοβούλιο σα είναι πάρα πολύ προσιλωμένο σε αυτό, στην πρόληψη. Αυτό είναι πραγματικά μια πράξη πρόληψης. Είναι μικρός, βραχής ο βίος συνήθως μιας ένοπλης σύραξης. Αλλά το Συμβούλιο Ασφαλείας επεμβαίνει αργά. Όταν, όταν κλιμακώνεται ε, μια σύραξη δεν κάνουμε αρκετά προληπτικά ε, ούτε μετά το τέλος της σύραξης για να αποφύγουμε ε, η μεταπολεμική περίοδος να γίνει προπολεμική μιας άλλης σύραξης την οποία δεν έχουμε δει αλλά στο παρελθόν είδαμε να επαναλαμβάνεται. Γίνεται ένας λόγος για τις μεταρρυθμίσεις των ΟΗΕ, των Συμβούλιο Ασφαλείας και παντού. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα σοβαρό πρόγραμμα για την πρόληψη, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, και να ε, ε, ε, εξυπηρετούμε ταυτόχρονα και τους τρεις στόχους, ειρήνη, ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα. Και το περιφερειακό επίσης. Είναι τέτοιος ο κόσμος σήμερα που μια εμπόλεμη ε, ζώνη η κατάσταση δεν αφορά μόνο την ίδια τη χώρα αλλά όλη την περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε και κυρία Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δώσατε. Θαυμάζω πάρα πολύ το έργο σας και ε, προσβλέπω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρους για την ειρήνη, την ανάπτυξη, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ahora vamos a empezar con, con el debate. Tenemos... τη Έχουμε ζητήσει μια σειρά συναδέλφων το λόγο. Έχουμε συγκεκριμένο χρόνο, άρα πάμε για τα δύο λεπτά μάξιμου. Και ο πρώτος που ζητήσει το λόγο είναι ο κύριος Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ελίασον. Θυμάμαι ότι είχατε εμπλαγεί με το Σύμφωνο Σταθός για την Ευρωπαϊκή Ευρώπη και και όσον αφορά την ασφάλεια επίσης και είχατε τότε πιο πολλές αρμοδιότητες. την Ουκρανία ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη έχει ασχοληθεί η διεθνή κοινότητα, αλλά όχι τόσο πολύ ο ΟΗΕ. Έγινε εκείνη η ορική ψηφοφορία πριν από ένα χρόνο, τότε που Γενική Συνέλευση ψήφισε υπέρ της καθικής ε, ακαιρεότητας. Ποτέ βέβαια δεν έχουμε ε, ομοφωνία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ε, λίγα περισσότερα για το πώς θα μπορούσε να εμπλακεί περισσότερο ο ΙΕ όσον αφορά την επίθεση κατά της Ουκρανίας. Και σχέση όλα αυτά που περιμένουμε για το μέλλον, γιατί επί τη βάση της εμπειρίας που έχουμε πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια συνολική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Κεραίρο Σαλόμ. Ευχαριστώ κύριε Λίασον για τα όλα όσα κάνετε και για το με πόσο δέμενο τρόπο μας παρουσιάσατε το τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους λαούς, τον κόσμο που χρειάζεται βοήθεια. Έχω δύο ερωτήσεις. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση τώρα τελευταία ούτω ώστε να κάνουμε κάτι για κάποιε ανθρωπιστικέ κρίσεις. Γιατί έχουμε ένα σωρό μείζονε κρίσεις στον κόσμο. Και διαπιστώνουμε ότι έχουμε περικοπές στα εμπιστιστικά προγράμματα και στεγαστικά προγράμματα. Για πέστε μας, ο ΙΕ τι μήνυμα θα μπορούσε να στείλει προς τα κράτη-μέλη και έτσι εκείνα να κάνουν κάτι. Οπότε να έχουμε μια παραπάνω χρηματοδότηση για συνολικές κρίσεις. Τώρα κάτι άλλο. Μιλήσατε για το πόσο σημαντικό είναι να επενδύσουμε σε κάποιο είδους αποδοτικά θεσμικά όργανα για αυτές τις μεταρρυθμίσεις που κάνετε στον ΟΗΕ όσον αφορά τα κριτήρια της διακυβέρνησης της δημοκρατικής υπέρ της σταθερότητας ούτω ώστε τα, να κάνουμε κάτι για αυτά τα αποτυχημένα κράτη, τα οποία είναι όλο ένα περισσότερα, και κάτι να κάνουμε πολέμηση φτώχεια και αποκλεισμού. Κυρία Έλιασον. Λέει κυρία Μπαστρίτσα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Λοιπόν, και πια πέστε μας γιατί έγινε για 22 ε, Ιανουαρίου, στη Γενική Συνέλευση του ΟΕ. Η πρόθεση ήταν να υπάρχει ένα πλαίσιο σε σχέση με τη χρήση του ίντερνετ για την διάδοση του φανατισμού, του μίσους κλπ. Επίσης τι λέτε για αυτό που είπατε ότι με τα ανθρώπινα δικαιώματα καταλαβαίνει ότι κάνει πάει στραβό όταν παραβιάζονται. Α, όμως τι γίνεται τώρα στη Βενεζουέλα. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά όμως εκεί έχουμε πολιτικές διώξεις, το έχουμε εμείς αυτό καταδικάσει και τι λέτε για την χρήση του στρατού, για την καταστολή. Και τώρα έχουν δεν έχουν τρόφιμα για πάνω από 40 μέρες εκεί. Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ηλίασεν για όσα μας είπατε. Και σαν προπαρασκευή για τη συνάντηση λάβουμε κάποια έγγραφα που αναφέρουν ότι θα μας ενημερώσει όσον αφορά το πώς έχουν τα πράγματα για την υλοποίηση του ψηφίσματος 1325. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ψήφισμα, αφορά ειρήνη και ασφάλεια. Και εκεί λέει ότι κάνετε μια μελέτη επιπτώσεων με θετικές διαπιστώσεις, αλλά όμως είπε η μελέτη ότι ο ΙΕ πόρο απέχει από το να μπορέσει να θέσει τέρμα στην βία μεταξύ των ΦΙΝΟΛ και επίσης για τα προβλήματα τα σχετικά με τις γυναίκες πρόσφυγες. Πεςτε μας δύο λόγια παραπάνω σχετικά αφορά αυτή τη μελέτη επιπτώσεων. Θα μπορούσε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Γκόμες, σας ε, βλέπω με μεγάλη χαρά και πάλι κύριε Λέσον και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε και αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πού βρισκόμαστε σήμερα τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εγώ θυμάμαι όταν εργαζόμουν εκεί ε, είχαμε μια ομάδα εργασίας ε, με ανοιχτή έκβαση αλλά ήταν μια ατέρμονη τελικά ομάδα εργασίας και πολύ σωστά τέθηκαν κάποια ζητήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει να αρχίσει αυτή η μεταρρύθμιση η Συρία είναι ένα ε, εύγλωτο ε, παράδειγμα πλήρους αδιεξόδου στο Συμβούλιο ε, Ασφαλείας με όλα τα συμπαρομαρτούντα της κρίσης αυτής. Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Δεύτερη. Συμφωνώ απολύτως μαζί σα για την Αφρική, για τις παράνομες εκροές οικονομικών πόρων, όπως είπατε, που είναι λόγω διαφθοράς. Κατά τα άλλα, όταν φεύγουν από την Αφρική, στι δικές μας τράπεζες καταλήγουν αυτά τα λεφτά στην Ευρώπη, έτσι. Τουλάχιστον αυτό λέει η έκθεση για τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα του περασμένου έτους. Και θα πρέπει και αυτό να το προωθήσει ο ΙΕ. Διότι όταν εμείς κοιτάμε και κοιτάξουμε ε, τις επιπτώσεις και ε, τα παρακλάδια του LuxLeaks ε, στο Λουξεμβούργο θα καταλήξουμε και σε αυτά και θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τους Αφρικανούς σε αυτή την προσπάθεια. Και ένα τελευταίο για την προσέγγιση που είπατε για την πρόληψη αναγνωρίζοντας την αποτυχία των Ηνωμένων Εθνών στη Σρι Λάγκα. Υπάρχει και η Λιβύη. Τεράστια ευθύνη φέρουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη στη Λιβύη πλήρης αποτυχία. Δεν κατάφεραν να γνωρίσουν ότι το βασικό ζήτημα των δομών ασφαλείας ήταν κάτι που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούσαμε να υποδιόμαστε ότι είναι πραγματικός ο στρατός και γνήσια αστυνομία στη Λιβύη όταν τίποτα από αυτό δεν συνέβαινε. Θα πρέπει να το καταλάβει Υπάρχουν κάποιοι που μας είναι ιδιαίτερα αγαπητοί και προσφυλείς για την ανθρωπιστική μας βοήθεια, αλλά ουσιαστικά είναι στιγμή δικτάτορες. Και κοιτάξτε τι γίνεται και στην Αιθιοπία που είναι και η αντίσταμπέμπα πρωτεύουσα της Αφρικανικής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ελίασον για την εμπνευσμένη σας παρέμβαση και ο ενθουσιασμό σας είναι κάτι που πραγματικά χρειαζόμαστε ε, στον δρόμο μας προς ένα καλύτερο κόσμο. Εδώ είμαι, αν δεν με βλέπετε. Επίσης γνωρίζω ότι παίξατε ρόλο κλειδί στην πρόθεση του κράτους δικαίου στο διεθνές πλαίσιο για την ε, αηφόρο ανάπτυξη και τους αναπτυξιακούς στόχους. Και θα ήθελα να μάθω πώς πήγε αυτή η προσπάθεια και ποιοι είναι οι καλοί και οι κακοί στις επιδόσεις εννοώ σε αυτή την περίπτωση. Το κράτος δικαίου είναι βεβαίως εκ των όνου κάνευ για τους στόχους της χιλιετίας, γιατί όλα αυτά που βλέπουμε, πολλά προβλήματα, έχουν να κάνουν με την έλλειψη κράτους δικαίου, έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη λογοδοσίας. Mm Πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε καλύτερα το κράτος δικαίου ε, στο μελλοντικό πλαίσιο της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σίγουρα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Ελιασόν για, τις, για την παρουσίασή σα. Μιλήσατε για τη συμπερίληψη και τη σημασία των θεσμών, συμφωνώ απόλυτα. Στο Παγκόσμιο Αναπτυξιακό Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών έχουμε έναν, έναν αναπτυξιακό στόχο για τις θεσμούς που δεν αποκλείουν, δεν περιθωριοποιούν κανέναν. Θα έλεγα αυτό να εφαρμόζεται καθ' ολοκληρία, όχι μόνο σε αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Και εδώ υπάρχει μια σημαντική πρόκληση, γιατί έχουμε επιφανή μέλη του ΟΗΕ, κάποιες αναδυόμενες οικονομίες που αναπτύχθηκαν οικονομικά, αλλά σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θεσμών που δεν αποκλείουν αλλά συμπεριλαμβάνουν, φαίνεται ότι παλινδρομούν. Ε, πώς ε, μπορείτε να αντιμετωπίσετε το θέμα, γιατί έχετε πολύ πλούσια εμπειρία. Πώς θα αναλάβει και πώς θα ανταπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση το Οργανισμό Συνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ κύριε Σπαντσέρη. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Τι γνώμη σας, παρακαλώ, για δύο γενικού χαρακτήρα θέματα. Πρώτα πρώτα αυτές οι πολιτικές, γεωπολιτικές αλλαγές, οι οποίες πάρα πολύ επηρέασαν τη, τη κοινωνία, την οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα και περιφερειακή κλίμακα εγώ να πούμε ότι είναι αναμφισβήτητο ότι πάρα πολλέ από αυτέ τι ε, συγκρούσει που έχουν τόσα προβλήματα είναι συνέπεια του ότι δεν υπάρχουν πια τα, τα παλιά σημεία αναφορά. Μέχρι το 89 είχαμε τι τις δύο υπερδυνάμει, κατόπιν μετά είχαμε τι ε, ΙΠΑ μόνο και τώρα λιγότερο λειτουργούν όπω τότε είπα οπότε δεν έχουμε τώρα κάποιο είδους ε, ε, υποκατάστατα σαν σημείο αναφοράς. Δεν είναι η Ευρώπη σήμερα και από ό,τι φαίνεται αυτό δεν είναι ούτε η αποστολή του ΟΗΕ. Και ε, επίσης θα πρέπει επομένως να δούμε πώς σε περιφερειακό επίπεδο θα αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Μια νέα ερμηνεία της παγκόσμιας ε, ε, κατάστασης. Οπότε να δούμε πώς μπορεί ο ΙΕ να βοηθήσει τόσο ώστε να βρεθούν κάποια νέα σημεία αναφοράς. Δεύτερη πολύ σύντομη σκέψη. Υπάρχει εδώ μια αντίφαση που θα πρέπει να δούμε τι θα την κάνουμε. Δηλαδή, ε, τα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Και πολλές φορές στο βωμό της ε, οικονομικής πρόοδου θυσιάζεται ε, υπόθεση των δικαιωμάτων. Και το κάνει αυτό και η Κίνα και η Ρωσία. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, ούτως ώστε να είμαστε συνεπείς σε όσα διακηρύσουμε για ανάπτυξη και οικονομία. Α, με την ευκαιρία αυτή μια ερωτησούλα που με απασχολεί και απασχολεί πολλού ιστορικού λόγους στην Ισπανία. Τι είναι η Δυτική Σαχάρα. Είναι εδώ να απεμπλέξουν το θέμα που έχει κολλήσει και να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του αυτοπροσδιορισμού <coughs> για να σταματήσει εκεί η κατάσταση που επικρατεί. Γι' αυτό διάθεσε λίγο πρόεδρος. Κύριε Σεβάγιος, ευχαριστώ. Είχα κάποιες ερωτήσεις για την πρόληψη, την πρόληψη των κρίσεων. Αλλά διαπίστωσα με χαρά ότι το αναφέρατε και από μόνο σας και αποτελεί σημαντικό τμήμα του έργου σας και ελπίζω στο μέλλον να αποκτήσει, όλο, να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί ακριβώς δεδομένου πληθώρα των συγκρούσεων που έχουμε, χαίρομαι που επικεντρώνεστε και στην πρόληψη. Μιλήσατε για την ομάδα υψηλού επίπεδου που ασχολείται ακριβώ με τα θέματα της πρόληψης, ώστε να αποτρέπουμε σε σχετικά πρόωρο στάδιο την ε, δημιουργία πρόσφορα εδάφους για τις κρίσεις. Γιατί όπως είπατε δεν έχουμε εναλλακτικό πλανήτη, δεν έχουμε δεύτερο πλανήτη. Ε, γίνεται μια κούρσα τώρα για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και των πόρων και με την ε, όξυνση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων τα προβλήματα αυτά θα γίνονται ακόμη δυνότερα γιατί αν δεν ε, βρούμε μια λύση θα χειροτερεύουν ε, οι κλιματικές αλλαγές. Πώς θα προστατεύσουμε στο μέλλον την Αρκτική. Γιατί για την Ανταρκτική έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο προστασία. Στην Αρκτική όμω πώ θα την προφυλάξουμε. Νομίζω ότι και αυτό το θέμα θα πρέπει να το θίξουμε. Κύριε, ο κύριο Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Έλιασον, και να πω ότι μιλήσατε μεταξύ άλλων και για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην ομιλία σας. Εγώ είμαι ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ακριβώς μετά το 2015. Μας είπατε κύριε Αναπληρωτή ε, Γενική Γραμματεύ ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ε, χειροπιαστούς αριθμούς και καλές λύσεις ε, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο μέλλον. Ερωτώ λοιπόν, τι θεωρούσατε ως επιτυχία της διάσκεψης της Αντισαμπέβα, ποιες θα ήταν καλές γιατί, ε, λύσεις, γιατί ο Ιούλιος ε, είναι πολύ κοντά. Οπότε, τι περιμένετε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό και ε, πώς κρίνετε τα σημάδια που δίνουν οι άλλοι βασικοί εταίροι και δωρητές της αναπτυξιακής βοήθειας και τι περιμένετε για να θεωρήσετε ότι είναι επιτυχημένη η μελλοντική αυτή διάσκεψη του Ιουλίου για το μέλλον της ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριος Μπούχνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λίασον αφού ήρθατε στο Κοινοβούλιο να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Θα ήθελα να επανέλθω λίγο στην δεκάτη επέτειο του ψηφίσματος 1325. Όπως θα γνωρίζετε σίγουρα, η κατάσταση ιδιαίτερα των γυναικών σε ορισμένες χώρες έχει επιδεινωθεί ικτρά το τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα να θυμίσω ότι κάθε μέρα εκατοντάδες κορίτσια και γυναίκε στα μίλ στη Σρι Λάνκα βιάζονται από στρατιωτικούς. Θυμίζω την κατάσταση στην Αίγυπτο, όπου αυξάνεται η βία κατά των γυναικών, ιδιαίτερα κατά των χριστιανών, που τις απαγάγουν ε, και τις μεταχειρίζονται, τις ε, ε, ζητούν λίτρα όταν δεν πληρώνονται τα λίτρα, τις σκοτώνουν και παίρνουν τα όργανα του για μεταμόσχευση. Η κατάσταση ε, φαίνεται να συναντά την ανοχή ε, της κυβέρνησης της Αιγύπτου. Δεν κάνουν τίποτα, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ενέχονται κιόλα. Εμείς ε, θα παραμείνουμε θεατές. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κάνουμε κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ετήρησαν τον χρόνο και θα δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Ελίασον για να απαντήσει με την ησυχία του στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω απολύτως στις ερωτήσεις σας, όλες πολύ σημαντικές. Ε, αλλιώς δεν θα <laughs> μπορούσατε να διπνήσετε αν ε, επεκτανθώ σε όλες τις ε, ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Ο ΙΕ δεν ενέχεται πολύ στην ουκρανική κρίση, τουλάχιστον όχι όσο θα θέλαμε. Τα προβλήματα ε, ισχύουν ε, ακόμα περισσότερο για την Ουκρανία τα ψηφίσματα, ενώ όπως αναφέρθηκε και στη Συρία. Στη Γενική Συνέλευση έγινε πολύ σημαντική ψηφοφορία όπου διατρανώθηκε ότι το θέμα της εδαφικής κεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων είναι σαφές ε, ήταν πάρα πολύ σαφές το μήνυμα και για το θέμα της Κρυμαίας. Ο Γενικός Γραμματέας και εγώ πάντα είμαστε διαθέσιμοι για να προσφέρουμε τις καλές υπηρεσίες μας. Ξέρετε ότι αρχές Μαρτίου πήγα στην Ουκρανία σε μια σημαντική στιγμή της κρίσης πριν τα γεγονότα της Κρυμαίας και ε, ο Γενικός Γραμματέας ήταν σε συχνή επαφή με την ηγεσία και της Ρωσίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας δηλαδή και της Ουκρανίας της ίδιας. Εμείς με χαρά να παίξουμε αυτό το ρόλο μας, αλλήμωνο, αν υπάρχει ανάγκη ε, βαροχής καλών υπηρεσιών που να το αναγνωρίζουν τα ενεχόμενα μέρη αλλά και άλλοι σημαντικοί πρωταγωνιστές. Είμαστε στη διάθεσή σας. Στο μεταξύ βεβαίω θα δραστηριοποιούμεθα στο ανθρωπιστικό μέτωπο που είναι ήδη τεράστια η πρόοδος και δυστυχώς αυξάνονται τα προβλήματα και ε, στην παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Είμαστε σε στενή συνεργασία και με τον ΟΑΣΕ στη Βιέννη. Αλλά εδώ φαίνονται και οι περιορισμοί στις ικανότητες και στη δράση που έχουμε σε ορισμένες καταστάσεις. Δεν έχουμε κοινή δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας και κατεύθυνση που να μας δίνεται. Η ανθρωπιστική κρίση καταλαμβάνει ένα τεράστιο τμήμα ε, και των προγραμμάτων και των ε, πόρων μας και των κρατών μελών αλλά και των Ηνωμένων Χαίρομαι πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας και θα ήλπιζα να μπορέσετε να στείλετε ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς τους ψηφοφόρους σας στις χώρες σας. Υπάρχουν τεράστια δεινά στο Λίβανο το Δεκέμβρη που πήγα τελευταία φορά. Το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα ε, άρχισε να δίνει συσίτια ε, στον κόσμο που χρειαζόταν φαΐ για την ημέρα. Με δελτία. Ευτυχώς καταφέραμε να σταματήσουμε πολύ γρήγορα αυτό το κίνδυνο, αλλά αυτό δείχνει πόσο ευάλωτοι είμαστε. Κάποτε ήμουν συντονιστής ε, επιγουσών καταστάσεων, σήμερα ο Βαλερία και τότε το 70% ε, των χρημάτων ε, τα απορροφούσαμε σήμερα 30 με 40% και είμαστε και ευχαριστημένοι. Είναι τεράστιες οι ανάγκες. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Συρία και την ίδια και τις γειτονικέ χώρες. 7 με 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι τεράστια ποσά αυτά. Και θα πρέπει να μπορούμε να κινητοποιούμε πόρους, αλλά και να βγούμε από την κατάσταση αυτή, να αντιμετωπίσουμε το κακό στη ρίζα του και να μην πέσουμε σε ε, αυτή την απέλπιδα ε, ε, αέναη διαιώνιση αυτής της κρίσης. Ένα δισεκατομμύριο χρειαζόμαστε και μόνο για να μένει ο κόσμος ζωντανός, αλλά θα πρέπει να γυρίσει στις αιστείες του, να κάνει μια κανονική ζωή. Πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται και αποκατάσταση. Αλλιώς είναι φαύλος κύκλος. Και οι δικοί σας οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι έχουν δυσκολίες να πληρώνουν αυτά τα τεράστια ποσά, τα θεώρητα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, για τους ε, καλούς θεσμούς και τη σωστή λειτουργία. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Και αναφέρατε κάτι που έχει να κάνει με τη σχέση μεταξύ καλών θεσμών και ε, ε, σταθερότητας. Πολύ σωστά είπατε. Μια χώρα που δεν έχει θεσμούς καθόλου, είναι πάρα πολύ αδύναμη ε, σε πολλούς τομείς, είναι μια ασθενής χώρα, μια ευάλωτη χώρα και πολλές φορές μια αποτυχημένη χώρα. Και όταν είσαι μια χώρα που αποτυχάνει ή έχει ήδη αποτύχει, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η χώρα αυτή. Γιατί εγκυμονούν κίνδυνοι ε, ταραχών, εμφυλίων πολέμων και περιφερειακών κρίσεων. Η καλύτερη λοιπόν συνεισφορά που έχει μια χώρα σήμερα να κάνει είναι να φροντίζει τους πολίτες τους ίδιους χωρίς αποκλεισμούς, με ισχυρούς θεσμούς που να εγγυώνται μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτό δεν είναι μόνο καλό για τον ίδιο το λαό μιας χώρας, αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια και ειρήνη τη σήμερα ημέρα. Εγώ θέλω να το δω και από την άλλη σκοπιά. Θα το πήγαινα τόσο μακριά λέγοντας ότι οι διεθνείς λύσεις για το κλίμα, για τη μετανάστευση, για αυτά τα παγκόσμια ζητήματα η καλή διεθνής λύση και φόρμουλα στο σημερινό κόσμο είναι προς όφελος των δικών μας, των ιδίων εθνικών συμφερόντων των κρατών μας. Αν υπάρξουν καλές διεθνείς λύσεις, αυτό συμφέρει και τις χώρες μας και την καθημερινή μας ζωή και τα εθνικά συμφέροντα κάθε χώρες. Θα μπορούσατε να φανταστείτε τι θα γινόταν στον κόσμο εάν όλα τα κοινοβούλια, οι αρθρογράφοι, και ο κόσμος έβγαινε στους δρόμους και έλεγε θέλουμε αυτή τη διεθνή συμφωνία γιατί είναι στο δικό μας εθνικό συμφέρον. Για να σπάσει αυτή η τεχνητή διάκριση μεταξύ εθνικού και διεθνού συμφέροντος. Αυτό χρειάζεται. Αυτό κάνετε κι εσείς άλλωστε εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Δεν μπορώ να μιλήσω για τα εγκλήματα μίσου στο διαδίκτυο. Δεν μπορώ να αποφανθώ γιατί δεν γνωρίζω πολύ καλά αυτό το θέμα μόνο ε, ακροθυγός. Ε, ε, είναι το κλασικό δίλημα η ελευθερία της έκφρασης από τη μια και από την άλλη ο σεβασμός των ε, παραδόσεων, των πολιτισμών και η μη υποδάβληση ακραίων αντιδράσεων. Αλλά δεν μπορώ να πω, δεν, δεν έχω γνώση καλή του θέματος για να το συζητήσω μαζί σου μαζί σας. Το ίδιο ισχύει και για τη Βενεζουέλα. Δεν παρακολουθώ την κατάσταση στη χώρα. Ναι, είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας εκλεγμένο ε, με πολλές ψήφους και είναι και ο κατεξοχήν υποψήφιος των ε, χωρών της Λατινικής Αμερικής. Σε σχέση και με συνέχεια όσο είπα προηγουμένως, δεν ε, διστάζουμε να στιγματίζουμε ε, της παραβιάσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είμαι πολύ περήφανος που μόλις ε, διορίσαμε τον Σαΐτ Χουσείνος νέο ε, είπα το αραπαστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γενέβη και είναι σαφέστατος και ίδιος στις δηλώσεις του. Και ελπίζω να συνεχίσει αυτό το δρόμο το Συμβούλιο Ασφαλείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είδατε πόσο αμαυρωθήκαμε. Είπα δεν θα κάνει τίποτα και τώρα έχουμε αυτούς τους ειδικού εισηγητές, έχουμε αυτές τις ε, ειδικέ διαδικασίες. Οπότε, α, τώρα ε, ο φόρης του ανθρωπινά δικαιώματα κάτι πάει να κάνει τώρα. Για το ψήφισμα, μην πείτε στη γυναίκα μου ότι ξέχασα να σας πω για το 13-25. Προσοχή, προσοχή όσοι σου ακούνε γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ειρήνευση, σταθεροποίηση της ειρήνης τέλος πάντων και είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε αυτή την συνεχή αναβιώρηση όχι μόνο των επιχειρήσεων των ειρηνευτικών, τώρα θα έχει προγραμματιστεί για άνοιξη ε, θέρος, αλλά έχουμε και την ε, αναθεώρηση συνόψη του, του 2025 και είπα, είπαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και εγώ έχω γίνει διαμεσολαβητή σε έξι πολέμους και ποτέ δεν είδα από την άλλη μεριά του τραπεζιού μία διαπραγματεύτρια. Πάντως, πάντοτε είχα εγώ γυναίκες μαζί μου και στον Ταρφούρ είχαμε 25 γυναίκες που ήταν παρατηρήτριες των διαπραγματεύσεων και στη Σύρτη βέβαια πολλές από αυτές την πλήρωσαν όταν γύρισαν, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ακόμα τεράστιο έργο που πρέπει να επιτελέσουμε και επίσης όπως είπαν άλλοι δεν είναι μόνο το θέμα του να συμμετέχει κανείς σε μια ερνευτική αποστολή, αλλά είναι και το θέμα της ε, βίας, της οργανωμένης, συστηματικής βίας που υφίστανται οι γυναίκες, το οποίο είναι όπλο πολέμου, κατά τέτοιο απεχθή τρόπο. Και τώρα για την τελευταία ερώτηση, από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάτι σαν ανταγωνισμός του ποιο θα είναι πιο απέσιος εν μέσω αυτών των ε, τρομοκρατικών ομάδων ο ένας πάει να ξεπεράσει τον άλλο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να θυμούμαστε ότι αυτό γίνεται επίτηδες. Επίτηδες για να δημιουργεί φόβο. Αυτές οι ομάδες θέλουν να φοβόμαστε. Θέλουν να είμαστε φοβισμένοι, νευρικοί, να, να, να βλέπουμε πώς μας παρακολουθεί, κάποιος μας απειλεί, κάποιος. Αυτό είναι η πρόθεσή τους, ούτω ώστε να συρρυκνώσουν την ε, αξία, την ομορφιά της δημοκρατικής μας κοινωνίας θέλουν να μας, κάνουμε, να να αντιδρούμε υπερβολικά και να αντιδρούμε με έναν τρόπο που δεν ε, συνάδει πως αυτή την κοινωνία που με ε, έχουμε οικοδομήσει να είναι μια πρόκληση μεταρρύθμιση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Α, τώρα με στριμώχνετε πολύ. Mm. Γιατί επειδή έχω δουλέψει στην ε, γραμματεία, πάρα πολύ δύσκολο να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Θα μπορούσα να το κάνω σαν πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Αλλά τώρα που είμαι αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, δεν μπορώ. πάντω να σα πω ότι η μεταρρύθμιση όντω χρειάζεται. Το χρειάζεται στο μέλλον το Συμβούλιο, το χρειάζεται σήμερα για να αποκτήσει μια νοημοποίηση, να είναι πιο αντιπροσωπευτικό από ό,τι σήμερα. Και αυτό μάλλον είναι γενικότερη παραδοχή όλων. Επίσης, θεωρώ ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει ε, εν ώψη των όσων γινόντουσαν στον που πολυβροφές δεν θέλουμε να ξαναέρθει να μην είναι μόνο ένα διαπραγματευτικό όργανο γιατί αν κανείς έχει αρνηση κυρία τότε αυτό είναι ένα δώρο από την ε, διεθνή κοινότητα. Ότι δηλαδή πέντε κράτη μπορούν να ασκούν βέτο. Αυτό είναι ένα δώρο, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι και μια ευθύνη ούτω ώστε να μπορεί κάποιο να ε, γίνεται πρωτοπόρο για εξέβρεση κοινή λύση. Και να μην γίνεται το βέτο αποτυχία όταν το χρησιμοποιεί κανεί, δηλαδή το χρησιμοποιεί κανεί, σαν εναλλακτική στο ότι δεν μπόρεσε να κάνει διαπραγματεύσει. Οπότε γι' αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το σύνδρομο του ψυχρού πολέμου το να αποδέχεται ω κάτι το φυσιολογικό την άσκηση του βέτο, την απειλή άσκηση του βέτο. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε σε διαπραγματεύσει να μην καταθέτουμε τα όπλα. Να έτσι, σαν αστιάκι, να σα πω κάτι σε σχέση με το, το Σύμβουλο ασφαλεία. Α, η Καθολική Εκκλησία τι κάνει όταν εκλέγει τον Πάπα. Δεν είναι κακό το ότι τους κλειδώνει τους ε, καρδινάλιους εκεί τη Σάντα Συστήνα και βγαίνουν μόνο όταν βγει ο Λευκός Καπνός, μόνο όταν τα καταφέρουν να εκλέξουν τον Πάπα. Να, αυτό είναι ενδιαφέρον σαν ε, ε, παράδειγμα προς μίμηση. Για να το κάνουμε ίσως κι εμείς. Τι είχαμε άλλο για τη χρηματοδότηση, τα είπαμε, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το κάνει, σας ευχαριστώ. Είναι ντροπή που 50 δις δολάρια φεύγουν από την ομοδοτήση της Αφρικής. Σας ευχαριστώ για την προσφορά βοήθειας. Τώρα για την πρόληψη, ναι. Η Λιβύα τώρα βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα έπρεπε προληπτικά. Εκ των προτέρων έχουμε κάνει πολλά. Πάντω ακόμα το πράγματα γίνουν χειρότερα. Έχουμε σημαντικέ συνομιλίε στην Γενέβη με τους εκπροσώπους και όλο ένα και περισσότεροι εμπλεκόμενοι μπαίνουν στο παιχνίδι. Αλλά τα πράγματα δυσκολεύουν ακριβώ γιατί έχουμε και κάποιες κινήσεις ακραίες. Οπότε κάνουν τα πράγματα δύσκολα αν όχι αδύνατα. Επίσης, ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να βοηθά όσον αφορά την υποχρέωση της προστασίας που έχουμε. Ακριβώς όπως αποφάσισε η Γενική Σύνδεση το 2005. Αυτό θα μας βοηθήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως είπα και στην αρχική μου ομιλία. Και τώρα είπαμε βέβαια για το κράτος δικαίου και τα σχετικά θεσμικά όργανα αλλά έχει τόσες πλευρές αυτό το ζήτημα να σας πενθυμίσω στις 25 Ενάτου του 12 υπήρχε μια πάρα πολύ ε, σημαντική συνάντηση υψηλού επίπεδου με 44 χώρες εκεί στο, στον Νοία στη Νέα Υόρκη που είπε ότι το κράτος δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση σε σχέση με το θεματολόγιο της ανάπτυξης και για την ε, ειρήνη και για την ασφάλεια και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε το σχετικό έγγραφο ε, θα πρέπει να το έχουμε Ευαγγέλιο γιατί τα καλύπτει όλα καταπολέμηση διαφθοράς, δικαιώματα ανηλίκων, δικαιώματα γυναικών, ένα άρτιο δικαϊκό σύστημα. Είναι απίστευτο. Να. Πρόκειται για εκατοντάδες εκατομμυρίων που είναι σαν να μην υπάρχουν. Γιατί δεν μπορούν να το αποδείξουν ότι υπάρχουν. Δεν μπορούν να ψηφίσουν. Δεν μπορούν να γραφτούν σε άλλη Δεν έχουν επιστοποιητικό γέννηση. Δεν υπάρχουν. Να, τι πάει να πει κράτο δικαίου. Γι' αυτό σας λέω ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω γιατί ε, το βλέπετε αυτό σαν την παραθεση βορρα βορρά-νότου. Μα είναι θέμα που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του να ζει κανεί σε τόσες περιπτώσεις και επίση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια των προσπαθειών. επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θεσμικά όργανα, τα σχετιζόμενα με το κράτο δικαίου. είναι το, το μέσο προς επίτευξη του σκοπού. Και ελπίζω ότι θα έχουμε πρόοδο με τη βοήθειά σας. Και από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα πρέπει να αναγνωριστεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ταυτόχρονα και οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Γιατί πολλοί σκέφτονται στην Αφρική, στην Λατινική Αμερική, ότι είναι μόνο θέμα πολιτικό τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, σημαντικό είναι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι στην παγκόσμια διακήρυξη Αυτά ονομάζονται και ως κοινωνικά, οικονομικά, εργατικά δικαιώματα. Άρα να το δούμε πραγματικά με την παγκόσμια διάσταση. Έτσι είναι ο κόσμος σήμερα. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι είναι θέμα βόρα-νότου αντιπαράθεση. Έχουν παγκόσμια χαρακτήρα αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ σημαντικό επίσης αυτό που είπατε για τον δύο στο διπολικό μονοπολικό κόσμο, περιφερειακό κατά ε, παγκόσμιο. Θα μπορούσαμε να τα λέμε μία ώρα πάνω σε αυτό. Όχι, μην το κάνουμε. Θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα σύμφωνα με τον οποίο θα αποδεχόμαστε τις ευθύνες μας σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε σε κάποια χώρα τοπικό επίπεδο, πολλές χώρες που δούμε σήμερα προβλήματα δεν, δεν καταπολεμούν την, την, την, τον αποκλεισμό ε, και έτσι δεν προστατεύουν ε, τις, κάποιου είδου δικαιώματα μειοψηφιών κλπ. Γιατί έχουμε λοιπόν τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο, το υπηρετικό επίπεδο όπω είσαι εδώ, αλλά έχουμε και το παγκόσμιο επίπεδο επίσης και να καταλάβουμε ότι αυτό κατά μείζωνα λόγο ισχύει για, τα, για τους χώρους και πρέπει να το εντοπίσουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα, από το παγκόσμιο μέχρι το τοπικό. Σε ένα τέτοιο κόσμο δεν μπορεί κανείς να διαφοροποιήσει τις διαστάσεις μεταξύ τους. Για ένα καλύτερο κόσμο θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι δική μας ευθύνη σε όλα τα επίπεδα. Δεν θέλω για να θεωρείται σαν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτό θα φόβιζε. Ο ΙΕ να είναι πρωτοπόρος και ταυτόχρονα ζητούμε από τα κράτη να είναι πρωτοπόρα. Αλλά μόνο εμείς, ο ΙΕ, σαν καταλήτης των ενεργειών των άλλων. Είπαμε. Χρηματοδότηση για ανάπτυξη. Ναι, αλλά δεν αρκούν οι παγκόσμιες τράπεζες. Χρειάζεται ο ιδιωτικό τομέας, χρειάζεται τι γίνεται στι χώρε. Να, έτσι να κινητοποιείται η χρηματοδότηση. Άρα, να, για το ρόλο μα. Α, τι, α, τελειώσανε αυτό, αυτό ήτανε. Α, τι πολύ, έχω κάνει και καθίσει στο πανεπιστήμιο, οπότε είδατε. Φλιαρό. Αλλά νομίζω ότι κάλυψα τις ερωτήσεις σας. Εκτός ίσως από κάτι που θα μου επιτρέψετε να σας ε, προσθέσω. Ή όχι, αλλιώς σταματώ εδώ. Ναι. Σας ευχαριστούμε κύριε Ελίασον. Λυπάμαι που σας διάκοψα έτσι, αλλά το έκανα για τους διερμηνείς. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε εγκαίρως, γιατί δουλεύουν πολλές ώρες στη συνεδρίαση. Πάντως νομίζω ότι μας κάνατε μια ευρύ επισκόπηση και δώσατε ε, διεξοδικές απαντήσεις ε, σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε συμπεράσματα, αλλά ε, ξεκινήσαμε το 2015 και μάλλον στραβά το ξεκινήσαμε στη διεθνή κοινότητα. Είδαμε τι έγινε στο Παρίσι με το ότι τη συνεχιζόμενη κρίση στη Συρία, τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ. Συνεχίζεται η κρίση ε, στο Κονγκό, στην Αφρική, στο Σουδάν, ε, ανθρωπιστική κρίση, έλλειψη πόρων, ε, προβληματική χρηματοδότηση, πολλές και διάφορες προκλήσεις. Πάντως, εσείς μας μεταφέρατε τουλάχιστον τη δική σας δέσμευση να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα και τη στράτευσή σας. Και είπατε ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά και τα συνδέσατε και με τους άλλους πυλώνες. Νομίζω το θέμα δεν είναι απλώς ένα ψήφισμα ή 17 στόχοι, ή 69 στόχοι. Το θέμα είναι κάποια βασικά στοιχειώδη πράγματα που κάνουν τη ζωή να αξίζει και να έχει ένα νόημα για να κάνουμε υποφερτή τη ζωή στον πλανήτη. Και νομίζω ότι αυτό το νόημα μας το μεταφέρατε πολύ καλά. Και μάλιστα είστε κάποιος που εκπροσωπεί την παγκόσμια κοινότητα και εκ μέρου τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τη Επιτροπή Ανάπτυξη και εκ μέρου των Ευρωβουλευτών θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμότητα που ήρθατε γιατί μα δώσατε πολύ σημαντικέ πληροφορίε για το έργο σα και προσβλέπουμε ε, σε περαιτέρω συνεργασία και με του συναδέλφου σα. Πάντω χαιρόμαστε για τι πολύ στενέ σχέσει και την επικοδομητική συνεργασία που έχουμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω στην έκτακτη συνεδρίαση που θα έχουμε σε 9 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή Εξωτερικών στις 7 το απόγευμα στο Στρασβούργο. Οι επόμενε είναι οι τακτικέ, 23 Φεβρουαρίου η πρώτη. Αλλά μην ξεχνάτε την έκτακτη στις, 7 ε, Φεβρουαρίου, στις 9 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο.